Right. Jean-Paul, are you? Right. No, uh, that, that, that's all right. Um, we've had about seven and a half. Γεια σας, περίπου 7,5 λεπτά ακαδημαϊκή περίοδος αναμονής. επιβραδύνουμε ώστε να μπορέσουν να φτάσουν και να ξεκινήσουμε έτσι σωστά. Έχουμε μια σύντομη μερίσια διάταξη σήμερα το πρωί γιατί κάποια πράγματα έχουν αναβληθεί. Αναβάλουμε λοιπόν την εξέταση τροπολογιών όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και τα λοιπά και τα οικονομικά σχετικά θέματα. Με αυτές τις αλλαγές γίνεται δεκτή ημερήσια διάταξη δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ευχαριστώ. Υιοθετείτε. Πρέπει να εγκρίνουμε επίση τα πρακτικά της συνεδρίασης της 2 Σεπτεμβρίου 2009. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει. Θεωρούμε ότι εγκρίνονται λοιπόν αυτά τα πρακτικά. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Όσοι ήθιστε και τώρα είμαστε και στο διαδίκτυο στη συνεδρίασή μας την κυρία Μάτα Αντρέσεν ε, από την ε, EFD θέλω να την καλωσορίσω αναπληρώτρια, αναπληρώνει τον κύριο Ρέστη Ρώση. Το χρονοδιάγραμμα για το 2010 της Επιτροπής μας θα το βρείτε στους φακέλους σας όπως υιοθετήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και όπως αναγγέλθηκε κιόλα και την προηγούμενη εβδομάδα θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη τώρα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ 21.00 μετά μεσημβρινή και ε, εγκαίρως θα σας ε, δοθούν οι λεπτομέρειες. Αυτό έγινε για να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεταφράσεις, ε, να υπάρχει η διερμηνία και όχι μόνο να δουλέψουμε στα αγγλικά. Και θα έχουμε ακόμα μια συνεδρίαση όσον αφορά τα θέματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Λοιπόν, εντάξει μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην εξέταση του θέματος που είναι πρώτο της έκθεσης του κυρίου Μπούλμαν όσον αφορά το σχέδιο του Συμβουλίου που τροποποιεί διατάξεις ε, όσον αφορά την οδηγία ΦΠΑ. Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή κύριο Μπούλμαν λοιπόν ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εδώ πρόκειται λοιπόν για διαβούλευση. Η διαβούλευση όμως ήδη ολοκληρώθηκε, έγινε από πλευράς μας στην έκθεσή μας που ομόφωνα εγκρίναμε στις 8 Ιουλίου 2008 από πλευρά συναδέλφου Ρωσάτη που είχε συνταχθεί από τον κύριο Ρωσάτη. Σε αυτή την έκθεση πρόκειται για το θέμα της ρύθμισης του ΦΠΑ όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμανσης, θερμότητας και την κοινή αντιμετώπιση επιχειρήσεων. Όλα αυτά δεν θέτουν προβλήματα. Πρόκειται όμως και για τους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος προκαταβολής ή ε, του ΦΠΑ όσον αφορά ε, πρώιμες καταβολές. Πρόκειται εδώ για μια απόφαση του Συμβουλίου που το πεδίο εφαρμογής το διευρύνει σημαντικά. Και έτσι δεν συνεισφέρει σε εναρμονισμό των φορολογικών θεμάτων αλλά εμβαλωματικά δημιουργείται ένα εμβαλωματικό έργο και σε σχέση με την εφαρμογή επεκτατικά αυτών των διατάξεων όποιος επιθυμεί μπορεί να το κάνει ζητήθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο μια και οδηγούμαστε σε σημαντικές αλλαγές εκ νέου να ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα και δεδομένη της πρότασης τώρα του Συμβουλίου που εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολική μπορεί κανείς πολλά θέματα στην προκαταβολή ΦΠΑ, στην αφαίρεση ΦΠΑ ε, σε σχέση με ακίνητα να τα δει. Η πρόταση δεν είναι απόλυτα σαφής, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν στην ενιαία εσωτερική αγορά και γι' αυτόν τον λόγο κάνω τις εξή προτάσεις που σας υποβάλλω. Πρώτα απ' όλα αποσαφήνιση που πρέπει να υπάρξει για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε κινητά τα οποία εντάσσονται ε, κινητές αξίες που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτών των ακινήτων. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το κοινό πλαίσιο ορισμού ώστε να μην έχουμε αυθαιρεσία από πλευρά των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, θέλουμε προτού υπάρξει διεύρυνση, επέκταση του πεδίου εφαρμογή εδώ, να γίνει μια εξέταση. Ποιε επιπτώσει θα υπάρξουν στην ενιαία εσωτερική αγορά, τι αναμένεται να γίνει σχετικά. Μια προεκτίμηση δηλαδή, προεκτίμηση της διεύρυνσης του πλαισίου για το πεδίο εφαρμογής. Διότι δεν επιθυμούμε, δεν θέλουμε να ε, ζημιωθεί, να ε, υπάρξει βλάβη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς με μια τέτοια διεύρυνση ή επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Και θέλουμε η εφαρμογή στον μηχανισμό διορθώσεως, δηλαδή αν υπάρχει υψηλότερη εκτίμηση σε ένα χρονικό διάστημα χ κάποιων οικοπαίδων, να υπάρξουν ρυθμίσεις και αποσαφηνήσεις, να μην καταλήξουμε σε αυθαίρετα δηλαδή πλαίσια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να επανέλθουμε να ξαναγυρίσουμε στην παλαιά σαφή ιδέα όπως είχε παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ρυθμίζει αυτό το θέμα να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη ας το πω έτσι πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και να μην έχουμε ε, προβλήματα και τρίβες που θα καταλήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή είναι η πρότασή μου και παρακαλώ λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας τώρα πλευρά σας. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λέει η Σε αυτή τη στιγμή δεν έχει ζητήσει κανεί ε, να πάρει το λόγο, δεν έχει κανένα ζητήσει το λόγο και εξάλλου δεν βλέπω και κανέναν σκιώδη εισηγητή. Ρωτώ λοιπόν την αίθουσα, θέλει κάποιο να πάρει το λόγο. Ναι, ε, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής φαίνεται ότι θέλει να μιλήσει και θα μπορούσαμε να τον ακούσουμε ενδεχομένω. Παρακαλώ πολύ. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά από τις εξηγήσεις που ακούσαμε, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας αν αποφασίσει να υπερψηφίσει την έκθεση αυτή και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον εισηγητή γιατί στήριξε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε πολύ απλούς ε, τρόπους ε, αναφερόμαστε στην αρχική ιδέα την οποία ε, είχαμε, δηλαδή να κάνουμε κάποιες μικρές τροπολογίες ε, τρέχον σύστημα, στο ισχύον σύστημα ΦΠΑ και συνήθως αναφερόμαστε σε αυτήν την τροποποίηση σαν τεχνικές διευκολύνσεις πρέπει να πω ότι υπάρχει μία πρόταση μείωσης μονάχα για τα ε, για τα έπιπλα και για ε, κινητές ε, αξίες. Αλλά βεβαίως η έκπτωση είναι δυνατή μονάχα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπάρχει η δυνατότητα αργότερα να διευρυνθεί προς κάθε είδους αγαθό χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε συγκεκριμένες περιοριστικές δράσεις. Ε, τώρα, σε γενικές γραμμές θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ε, να ε, του πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο την στάση... Αυτή την έκθεση και με την έκθεσή σας να σας επισύρω την προσοχή εις ένα. Ένα στοιχείο για να σας εξηγήσω την θέση μας. Μιλώ για την αιτιολογικη παραγραφω παραγράφο 10α. Which in our analysis... Κατά την δική μας ανάλυση η ουσία είναι ότι ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω πολιτική δράση. Κάτι το οποίο αφορά κάποια νομοπαρασκευαστική διαδικασία, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ σε μια τελική παράγραφο οδηγίας. Επί της ουσίας, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όσον αφορά θετικά ή αρνητικά για να δεσμευτούμε όσον αφορά τέτοιες περαιτέρω ενέργειες. Εδώ σταματώ για λίγο. Να ακούσουμε τον εισηγητή και αν έχετε τίποτε περαιτέρω απορίες είμαστε στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε και ξαναγυρίζουμε στον εισηγητή μια που άλλος δεν έχει στήσει το λόγο. Και θα πρέπει να σας τονίσω ότι στο παρελθόν αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι το να ε, υπάρχουν δίκαιο ανταγωνισμού και ισότητα στις επιχειρήσεις της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον ΦΠΑ και γενικότερα την ε, φορολογία. Αυτό το έχουμε ε, διατυπώσει με και στην προηγούμενη ε, θητεία. Ας επανέλθουμε επομένω στον κύριο Σιγητή. Ευχαριστώ για το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το σημείο που προαναφέρθηκε για άλλη μια φορά διμερώς θα το συζητήσουμε. Και Πρόεδρε, απομένει να πω κάτι ακόμα. Φυσικά στην αρχή της νέας κοινοβουλευτικής θητείας έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, πίεση δουλειά. Δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει χωρίς τις ε, εξαιρετικές εργασίες των υπηρεσία της υπηρεσίας μας της Γραμματείας. Ευχαριστώ γι' αυτό. Yes, thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Είναι περίεργο που το ξανά έχουμε τώρα το θέμα αυτό και πρέπει να ξαναδουλέψουμε με ταχύτητα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να περάσουμε στην επόμενη έκθεση σχετικά Μάλλον όχι, μάλλον όχι. Πρέπει να επανέλθω, λέει η Πρόεδρος. Η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 14η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Την 9η Νοεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες έτσι ώστε να ψηφιστούν στις 10 <coughs> Νοεμβρίου. Με την ελπίδα ότι ε, θα έχουμε την δυνατότητα να το ψηφίσουμε στον Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου. Από ό,τι βλέπω ο εισηγητής δεν έχει πρόβλημα και επομένως τώρα όντως μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2008. Η Εισηγητής ε, για το θέμα αυτό είναι ο Έντουαρτ Σικλούνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να αναφέρω είναι οι προθεσμίες. 20 Οκτωβρίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το προσχέδιο με την δυνατότητα να ε, κερδίσουμε μερικές μέρες, αλλά παρόλα αυτά τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στον Απρίλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν έχουμε καμία δυνατότητα, δεν μπορούμε να ε, καθυστερήσουμε άλλο. Ε, βεβαίως ε, είχα διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ε, Γραμματεία, είχα αρκετές συναντήσεις μαζί τους. Το ένα ζήτημα που υπάρχει είναι γιατί καταλαβαίνετε ότι η έκθεση αφορά το 2008 και πολλά πράγματα συνέβησαν το Δεκέμβριο του 2008 ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ε, αναλαμβάνουμε να παρακολουθήσουμε κατά κάποιο τρόπο όλα τα σημεία τα οποία ε, θίγονται στην έκθεση του 2008 και επομένως να, το να τα προχωρήσουμε μέχρι το 2009. Από την άλλη πλευρά επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να ε, έχω την δυνατότητα να ε, μετακινήσω κατά κάποιο τρόπο κάποιες τροπολογίες από την μία περιοχή της έκθεσης σε μία άλλη και ελπίζω ότι όσο προχωράμε θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε και τις τροπολογίες και τα θέματα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για το θέμα αυτό τώρα. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπάουτ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι. ναι. Οι προθεσμίες, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σφιχτές. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ε, τις εκλογές δεν ε, έχουμε καμία, κανένα περιθώριο. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί έκθεση για τον, να για τον Οκτώβρη. Βλέπουμε πάντως ήδη τον αντίκτυπο της κρίσης. Εάν λάβει κανείς υπόψη του την κατάσταση αναχώρα, διαπιστώνει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης είναι σαφής. Βλέπουμε εδώ ότι υπήρξαν τέσσερα δις αποθεματικό και περιμένω με ανυπομονησία τις ε, συζητήσεις ε, οι οποίες θα λάβουν χώρα τις επόμενες, τρει τις επόμενες τρεις εβδομάδες και είναι για να δούμε πού θα καταλήξουμε με τον εισηγητή. Πρόεδρος, δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητά το λόγο, κανένας από τους σκιώδεις εισηγητές, επομένως πολύ ωραία. Μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει παρότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό και δύσκολο να το σεβαστούμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, την 25η Μαρτίου ο κύριος Τρισέ έχει ήδη συμφωνήσει να είναι ε, μαζί μας και επομένως ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει υποβληθεί η δικιά μας, τα δικά μας σχόλια για την ετήσια έκθεση και επομένως αυτή είναι η τελική ημερομηνία και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και μια καλή έκθεση Λοιπόν, 9η Νοεμβρίου το προσχέδιο και 30η Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών έτσι ώστε να υπάρχει κάποια ε, χρονική δυνατότητα ενσωμάτωσης των τροπολογιών. Και είπαμε λοιπόν 27 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και 25 Μαρτίου Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 8. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Έχουμε έγγραφο εργασίας από τον εισηγητή, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Ε, έχετε το λόγο λοιπόν κύριε εισηγητά, κύριε Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για δεύτερη φορά λοιπόν αναφερόμαστε στην έκθεση αυτή για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Στα έγγραφά σας έχετε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο εκπονήθηκε με τις υπηρεσίες έτσι ώστε να υποβληθούν όχι ακριβώς λύσεις αλλά σημεία σκέψης δεν πρόκειται να αναλύσω εκ νέου αυτό το έγγραφο εργασίας το οποίο έχετε ήδη αναγνώσει, αλλά θα περιμένω σήμερα σχόλια, θέσεις δικές σας επί των διαφόρων θεμάτων ε, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια της συζήτησης για την οδηγία αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων για τις παρατηρήσεις σας. Um, Ο κύριος Κλίντς Frau Κυρία Πρόεδρε, διαβάσαμε λοιπόν το έγγραφο εργασίας ε, και είχαμε και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά από τότε τα πράγματα προχώρησαν κάπως όμως ε, δεν έχουμε ολοκληρώσει το δρόμο μας γιατί δεν έχουμε ακόμα την ίδια την έκθεση από πλευράς του εισηγητού. Διαπιστώνω όμως το εξής. Κατανοώ πλήρως ότι οι περιού λόγος ε, ε, διαχειριστές θέλουν, επιθυμούν τη συζήτηση. Όμως πρέπει να ομολογήσω ότι με λίγο από την επιμονή να γίνουν τόσες πολλές συζητήσεις μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. φαίνεται ε, ότι πολλές μετακινήσεις έγιναν μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Δεν έχει καμία έννοια να, μας, ε, να έρχονται και να μας λένε πράγματα γιατί συνήθως μας λένε τα ίδια πράγματα. <clears throat> Και από την άλλη πλευρά οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για το θέμα αυτό δεν είναι ε, μεγάλοι και άλλωστε και οι διαχειριστές που είδαμε δεν είναι και οι πιο σημαντικοί ε, διαχειριστές ε, Και πρέπει να πω επίσης ε, ότι ε, τα θεσμικά, οι θεσμικοί πόροι είναι περίπου του 47% ε, και τα property funds είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικοί πόροι και δεν εκπροσωπούνται ιδιαίτερως εδώ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να μην βρισκόμαστε βρισκόμαστε σε ομοιρία από μία κατηγορία ε, και όχι από ε, κάποια άλλη, δηλαδή να μην έχουμε τη δυνατότητα να ε, διευρύνουμε τη συζήτησή μας. από την άλλη πλευρά μια προσέγγιση που θα είναι ε, ίδια για όλους τους διαχειριστές μπορεί τελικά να είναι προβληματική. Εν πάση περιπτώσει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα τελικό έγγραφο που θα είναι χρήσιμο. Για να είναι χρήσιμο όμως χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Το έγγραφο το οποίο έχουμε μπροστά μας σαν έγγραφο θα πρέπει να τροποποιηθεί λέγω έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Όμως νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και η αντίδρασή μου είναι ότι ενδεχομένως θα πρέπει να, το ξαναστείλουμε στην, το σύνολο του θέματος στην Επιτροπή και να ξαναρχίσουμε από το μηδέν, αλλά δυστυχώς αυτό πια δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Ε, οπότε πρέπει κάποια στοιχεία να τροποποιηθούν. Τα κατόφλια, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν. γιατί θέτουν προβλήματα. Πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας. Ε, υπάρχει βεβαίως και το πρόβλημα των τρίτων χωρών. Αυτή είναι μια, ε, ε, καλή, ε, ένα, ένα μεγάλο πρόβλημα και τα depositories επίσης είναι ένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι σαν νομοθετική αρχή θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οδηγία αυτή όταν θα έχει ε, υιοθετηθεί θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς πρόβλημα. Και θα πρέπει λοιπόν να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε να είναι ε, αρμονικά συνδεδεμένοι με άλλες υφιστάμενες και ισχύουσες ε, οδηγίες. Ε, και ότι βεβαίως ε, δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τον ε, κατάλογο διαφάνειας κτλ. λοιπά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να επιτρέψουμε διπλή ή αντιτιθέμενη νομοθεσία θα πρέπει να μπορούμε να περάσουμε από την μία οδηγία στην άλλη, από το ένα νομοθετικό κείμενο στο άλλο, χωρί να υπάρχει καμία αντίφαση και καμία ασάφεια. Επομένω, το πιο σημαντικό είναι αυτός ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν να μην τον ε, ε, βάλουμε στη γωνία και να μην τον χτυπήσουμε περισσότερο. Επίσης δεν πρέπει η νέα οδηγία να καταστρέψει πράγματα τα οποία έχουν δουλέψει καλά μέχρι τώρα. Μπορούν και τα μεν και τα δε να λειτουργήσουν. Όσον αφορά τις ε, τρίτες χώρες, το πρόβλημα των τρίτων χωρών ενδεχομένως ε, θα λυθεί ευκολότερα εάν ε, διατηρήσουμε αυτά τα υφιστάμενα καθεστώτα. Τώρα, καθαρά για τις τρίτες χώρες. Στόχος μας πρέπει να είναι να βρεθεί λύση η οποία αφενός θα επιτρέπει όπως και στα OPSVM ε, να δημιουργούνται IFM ε, που θα έχουν κάποια σφραγίδα ποιότητος. Αλλά βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε φρούριο, δηλαδή να μην αφήνουμε τίποτα να μπει από πλευράς των άλλων χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το χειρό Ευρώπη. Θα πρέπει πάση θυσία να διατηρήσουμε την αρχή ότι η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή αγορά. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, ε, δημιουργούμε αδιέξοδα ε, για τους IFM και τους διαχειριστές IAF. Και θα πρέπει οπουδήποτε στον κόσμο βάσει των εθνικών αρχών να ε, υπάρχει δυνατότητα να πουλήσει κανείς στην Ευρώπη και η Ευρώπη βάσει ενός θεσμοθετημένου συστήματος να μπορεί να επενδύσει ε, στις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως που πρέπει να ρυθμιστούν. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ε, διαχειριστές που ε, είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη και που θέλουν ε, όμως να δώσουν ε, ας πούμε να κάνουν επενδύσεις με χρήματα, με πόρους που βρίσκονται εκτός Ευρώπης ας πούμε στα νησιά Κέιμαν. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς άδεια γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύπτεται από το ευρωπαϊκό ε, καθεστώς και βεβαίως ε, οι πόροι που βρίσκονται σε offshore εταιρείες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ε, έχουν αντιστοιχίες στην Ευρώπη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα αντιστοιχιών είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ περιμένω από τον εισηγητή προτάσεις συγκεκριμένα συγκεκριμένη για να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να γίνει ε, φρούριο, δεν μπορεί να ζητήσουμε τρία χρόνια για ε, μεταβατική περίοδο. Την τελευταία φορά είχα πει ότι προτιμούσα να, έχουμε, να περιμένουμε να έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάση ε, της έρευνας Σεζάρ για να δούμε τι θα κάνουμε με τις ΟΠΕΣΕΒΕΜ. Γιατί δεν είναι δυνατόν για τους θεσμικούς επενδυτές να έχουμε πιο αυστηρές διατάξεις ε, για, από αυτές που ισχύουν για τους τοπικούς επενδυτές. Η πρόταση της Επιτροπής είναι όχι μονάχα να υπάρχει ένα αρχείο για τους, και ένας κωδικός για τους ε, επενδυτές IFM αλλά και για τους άλλους διαχειριστές εναλλακτικών ε, ε, χαρτοφυλακίων και επενδύσεων. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει και το θέμα των παραβόλων θα πρέπει να το αφήσουμε γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και από την, εποχή, από την περίπτωση Μάντοφ καταλάβαμε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και επομένως θα πρέπει να βρούμε μια λύση που θα ισχύει και για τους IFM και για τους OPCVM. Επίσης, η εποπτεία και ο έλεγχος και ε, νομίζω ότι και η οδηγία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη και τις νέες διατάξεις ε, οι οποίες θα αφορούν την εποπτεία. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Βλέπω την αίθουσα για προσπαθώ να ζητήσω κάποιον σκιώδη συγητή και ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συμπαθάτε με συνάδελφο που δεν ήρθα στην αρχή της ε, συζήτησης ε, γιατί πλάνο ήρθα κατευθείαν από το από το αεροδρόμιο, είδα και άλλους αδέλφους που τρέχαν να προλάβουν. Θα πρέπει να συζητήσουμε, να συζητήσουμε με ψηφοφόρους, να συζητήσουμε με εταιρείε, με όλους τους θυγόμενους από αυτή την οδηγία, το σχέδιο οδηγίας και δεν μιλώ για τους συνήθεις ύποπτους. Γιατί εν προκειμένου σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων έχουμε θέματα και να δούμε τι γίνεται, ιδίως όσον αφορά τις ε, τρίτες χώρες, τι ισχύει όσον αφορά τις ισχύουσες ήδη οδηγίες για, αυτούς τους, για αυτά τα, τα, τα κεφάλαια, να δούμε τι ισχύει και τι πρέπει να γίνει. Έχουμε και το θέμα των συνταξιδοτικών ταμείων. Μίλησα με κάποιον διοικητικό παράγοντα της προάλλας αυτός διαχειρίζεται τους πόρους ε, ενός συνδικάτου. Μου και κοίτα να δεις, είμαστε αντίπαλοι πολιτικά. Αλλά με προβληματίζει αυτό το οποίο γίνεται, γιατί έχω χιλιάδες συνταξιούχους ε, στο δικό μου ταμείο και θέλω κάποια ευηλιξία ούτως ώστε να μπορέσω να έχω διαθέσιμα, διαθέσιμους πόρους παντού και στην Ένωση και εκτός ούτως ώστε να μπορώ να έχω την μέγιστη απόδοση για τους δεξιούς γιατί αυτοί αποταμιεύουν όλη τους τη ζωή και δεν μπορώ μια μέρα να γυρίσω για να τους πω έχω περιορισμού, ζορίζομαι κλπ. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τα hedge funds. Ξέρω ότι είναι διαβόητα, υπάρχουν κάποιοι φόβοι, όμως πάρα πολλές φορές είναι αποδοτικά. Άρα να κάτσουμε και να ζυγίσουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ε, οδηγίας για όλους. Τώρα, όσον αφορά τους συνταξιούχους. Προσοχή, εδώ υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα που μας περιμένει. Ε, γιατί ο μέσο ζωής ανεβαίνει, αυξάνει, τα παιδιά μας μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 100, άρα τους ταξιούχους να τους δώσουμε τα μέσα τόσο ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη μεγίστη απόδοση για τις ε, ποταμιές τους, για τις εισφορές τους. Κάτι άλλο τώρα Μίλαγα και με έναν διευθυντή ε, ξενοδοχείου και μου έλεγε για τα προβλήματα που έχει η αλυσία των ξενοδοχείων που δουλεύει, ανησυχούν για τη δουλειά τους, αυτοί που δουλεύουν εκεί ε, και τελικά μέσω κάποιου δανείου από κάποιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό όχι μόνο εξασφαλίστηκε το μέλλον της εταιρείας αλλά τώρα είναι και ρόδινο το μέλλον. επεκτάθηκε η αλυσία των ξενοδοχείων και δημιούργησε θέσει εργασία ακριβώ διότι αυτό το, αυτός ο οργανισμό, το Private Equity Fund, παρενέβη για να βοηθήσει. Μίλησα και με κάποιον πράσινο, Γερμανό, επενδυτή. Αυτός φτιάχνει τουρμπινοκινητήρε, χρησιμοποιεί την αιωλική ενέργεια και είπε ότι οι τράπεζε δεν μου δανείζουν και πάω σε κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου να δανειστώ. Venture capitals. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν από τη μια μεριά ζητάει να υπάρξουν περισσότερε επενδύσει και από την άλλη μεριά όμω δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο ε, στρέφονται προς μορφές που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει οι επιχειρηματίε και κυρίω αυτοί που βοηθάνε το περιβάλλον να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και προσοχή γιατί πολλέ φορέ αυτά τα κεφάλαια δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά στα οποία τελικά μπορούν να έχουν πρόσβαση οι επιχειρηματίε. Κάτι άλλο τώρα. Κάποιες επενδύσεις ε, για να βοηθήσουμε την παιδεία στην Αφρική. οι Ευρωπαίοι επενδυτέ, όπως έχει σήμερα η νομοθεσία θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο δηλαδή να πάνε στην ε, Αφρική και να επενδύσουν χτίζοντα κάποια σχολεία και αυτό να γίνεται απαρακόλλητα χωρίς εγγραφειοκρατίε. να κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό δούμε τι γίνεται άλλοι από τα νησιά Καϊμάνια θα την βρήκαμε και είπανε ότι προσπαθούμε σκληρά, δεν θέλουμε να είμαστε μια παραδοσιακή χώρα της Καραϊβικής και να ασχολούμαστε με μπανάνες, ρούμι και ζάχαρη και τέτοια εμπορεύματα. Θα πρέπει όντως να κάνουμε κάτι άλλο, να ασχοληθούμε με τις υπηρεσίες, τις χρηματοοικονομικές. Γιατί τα χρήματα που είναι εκεί έχουν αντίκρισμα. Μετράνε. Πέστε μας επομένως πώς θα μπορέσουμε να έχουμε απόδοση. Και μη μας βάλετε με μεταβατικές περίοδους και τριετίε. Τώρα πέστε μας τι να κάνουμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και κάτι έναντι αυτών των χρημάτων που έχουν βρεθεί εδώ. Για να βγει ο Κοσμάκης από τη φτώχεια. Τελευταίο τώρα σημείο που θέλω να πω είναι αυτό που αφορά τον κίνδυνο, τη διακινδύνευση. Ε, και εδώ τώρα λίγο θα το περιαυτολογήσω. Ασχολήθηκα με την επιστήμη των συστημάτων, έκανα και ένα διδακτορικό για συστήματα. Όλα τα συστήματα, οικονομικά, πολιτικά, όλα θα με απασχόλησαν και ε, επομένω σπούδασα την συστημική ανάλυση σε σχέση με ε, αυτή την οδηγία. Επομένω, ξέρω το, κάτι το οποίο με, με, με, με, με, φοβίζει. Ε, αυτό για τι καταθέσει. Πόσε είναι οι τράπεζε που σήμερα με αυτή την οδηγία θα μπορέσουν να, να είναι οι θεματοφύλακε που προβλέπετε εδώ Τέσσερις, έξι, πόσες τράπεζες. Για πέστε μου, πόσοι. Έξι τέτοιοι θεματοφύλακες θα είναι. Και όσον αφορά την ευθύνη, αυτά, ε, αυτές οι τέσσερις έξι τράπεζες θα έχουν περιόριστη ευθύνη, όμως αυτό συστημικά είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε και ποιε θα είναι οι συνέπειε. Τώρα για τη μεταδοτική περίοδο είναι κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Εάν τώρα βλέπουμε τα κριτήρια, γιατί να περιμένουμε τρία χρόνια. Να του δώσουμε κάποια, κάποια περιθώρια, κάποια δικαιώματα. Grandfather rights. Κάποιοι λένε για δεκαετία. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται κάποια κυκλική εναλλαγή. Άρα, για να δούμε προσοχή γιατί αυτό το θέμα αφορά όλη την Ευρώπη, όλους τους ψηφοφόρους. Άρα αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Καμάρα. Οι σκιώδεις εισηγητές πρώτα που θα ακούσουμε. Επόμενος, ο κύριος Καντήλ παρακαλώ. 11 η ώρα να το δίνετε λέει απόψε, οπότε και εγώ μόλις τώρα μπόρεσα να έρθω. Και καλύτερα να τηρείτε το πρόγραμμα το οποίο προβλέπετε. Αν θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων που να αποδίδει κάτι. Η πράσινη, όσον αφορά την οδηγία, να σας πω τι άποψη έχουν. Πρώτον, όσον αφορά το κατόφλι. Θεωρούμε ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα υπάρχει ε, ένα κίνδυνος γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρακαμφθεί αυτή η οδηγία από κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια τα οποία να διαβρώσουν το σύστημα. Άρα δεν θα πρέπει κατά τη να υπάρχει κάποιο είδου κατόφλι και θα πρέπει το σύνολο των πόρων, των κεφαλαίων να καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Και αυτά τα λέμε έχοντας επίγνωση του ότι υπάρχουν ε, κάποιες διατάξεις που θα πρέπει να θεσπιστούν όσον αφορά τα private equities. Γιατί ακριβώς δεν, έχουν, δεν, δεν, δεν διέπονται τα πάντα από τους ίδιους κανόνες του ίδιο πνεύμα. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή, Ρυθμιστική Αρχή. Εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει τα κεφάλαια εκείνα τα οποία έχουν κάποιο είδους ευρωπαϊκό διαβατήριο, αυτό το διαβατήριο να τους χορηγείται όχι από εθνικές αρχές, αλλά από κάποια πανευρωπαϊκή αρχή. Διότι θεωρούμε ότι εδώ ελοχεύει πραγματικό ε, κίνδυνο ανταγωνισμού μεταξύ των εθνικών αρχών. Και αυτό μπορεί να μα οδηγήσει σε κάποιο είδου ε, θεσμοποιημένη διαιτησία που θα κατεβάσει τον πύχη, θα μειώσει την ωφέλεια από αυτήν την οδηγία. Σε αυτή την οδηγία έχουμε ενσωματώσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, κάποια στοιχεία τα οποία τα έχει συζητήσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή τη δέσμη μέτρων για να καταλήξουμε σε κάποια πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Επομένω, αυτού του είδου η πιστοποίηση, αυτό το διαβατήριο ε, να δίνεται από κάποια από αυτέ τι πνευροπαϊκέ αρχέ που θα δεσμευτούν από αυτή την οδηγία. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά αυτό το υπομόχλιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα που να περιορίζει. Δεν υπάρχει κάποιο νούμερο, κάποιο όριο το οποίο να περιορίζει το πώς είναι δυνατόν να έχουμε ε, κάποιο τέτοιο υπομόχλιο για τα hedge funds. Όμως, όταν έχετε η κρίση, μπορεί να προβλέπει κάποια τέτοια εξαίρεση και με αυτό προβλέπεται να το κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προβλήματα όμως είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μονίμως ε, κάποιο τέτοιο μέσο παρέμβασης και όχι μόνο σε περίοδους κρίσης. Και πριν την κρίση ακριβώς για να προλάβει κανείς την, την, την, την επίθεση από την κρίση. Οπότε είμαστε υπέρ του να θεσπιστεί κάποιο ποσό ε, το οποίο να αφορά μέσω όρο ε, ανατρίμηνο, ανεξάμηνο και έτσι να μπορεί να περιορίσει αυτό, αυτό το είδος τα κερδοσκοπικά κεφάλαια. Επίσης, ε, να, να, μην είναι μόνη αρμοδία κομισιών, αλλά να εισαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά την αμοιβή, την αποζημίωση, για το οποίο τίποτα δεν, καθόλου δεν ρυθμίζει αυτή η οδηγία, ε, θα πρέπει να προβλέπετε κάποιο, κάποιο ελάχιστο θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο ε, συζητήθηκε στο G20 με το πόνους μάλους όσον αφορά αυτήν την ε, αντιστάθμιση, όσον αφορά αυτήν την αμοιβή, ούτως ώστε να μπορούμε να αντισταθμίσουμε το ρίσκο από τα hedge funds. Και θα κάνουμε αυτό το οποίο ελέγχθη στο G20. Κάτι άλλο. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα των τρίτων χωρών. Είμαστε μάλλον υπέρ της αρχής της ισοδυναμίας. Αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κάποιο δίκαιο και αυτό να εξάγεται και κατόπιν. Να παρασύρονται προ τα πάνω οι υπόλοιπε χώρε τόσο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στι αγορέ μα, τότε πάμε προς τη κατεύθυνση. Πάντω, επιφυλασσόμαστε πάρα πολύ όσον αφορά τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, διότι έχει να αντιμετωπίσει κάποιε πιέσει που θα ασκήσουν κάποιε χώρε. Χώρε που θα θεωρήσουν ότι ένα τέτοιο ρυθμιστικό πλαίσιο ε, είναι τέτοιο που αντιβαίνει στο δικό του ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένω, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το συζητάει και το Συμβούλιο. Άρα, εμεί θέλουμε καταρχήν να ισχύσει η αρχή τη οδυναμία και να ενισχυθεί. Και έτσι να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότεροι παράγοντες αντικειμενική και να μην υπάρχει τόσο ευρύ περιθώριο ελιγμών και περιθώριο ερμηνεία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο στην οδηγία, τότε να υπάρχει κάποια ρύθμιση πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά τα hedge funds στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία ε, είναι offshore και λειτουργούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούμε ότι μια τέτοια αυτή ρύθμιση δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ήδη ο ΠΟΕ λέει ότι εάν και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αντιστοιχεί στις ανάγκες αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων είναι κάτι το επιτρεπόμενο. Επομένω, δεν έχουμε εδώ πέρα κάποιο είδου ε, σύγκρουση με τι διατάξει του ΠΟΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω αισθανόμαι ότι θα έπρεπε να αντιδράσω και να απαντήσω στο θέμα του συντονισμού του χρονικού με τον τρόπο που πάντα προηγούμενα υιοθετεί το, χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικού χαρακτήρα φυσικά και η συζήτηση για ένα θέμα αν δεν είναι ιδιαίτερα ας το πω έτσι χρονοβόρα αλλά επισπεύδονται άλλα θέματα και είναι ατυχές σε σχέση με τους σκιώδεις εισηγητές για τα δύο προηγούμενα θέματα που δεν βρισκόντουσαν είτε δεν βρισκόντουσαν εδώ είτε δεν είχαν ζητήσει τον λόγο να παρέμβουν και έτσι είχαμε σύντομη συζήτηση. Αυτό σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα συνεχίσουμε με αυτή τη συζήτηση. Έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο και ελπίζω ότι τα μέλη θα αισθάνονται ότι προσθέτει αυτό στην ποιότητα της συζήτησης. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ούντο Μπούλμαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το χρονοδιάγραμμα προφανώς και τον δικό μας και τον κύριο Γκόμπετς, τον παρακόλλησε να, να παρέμβει. Μπορώ όμω όλου να του καθησυχάσω. Νομίζω η νομοθεσία στην πρώτη συζήτηση αυτή δεν ρυθμίζεται τελεσίδικα, αλλά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων από την εργασία τη εργασία αυτή τη Ευρωβουλή μα. Τώρα για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα την εικόνα της φυλακής να ξανααναφέρω που από πλευρά σας συναδέλφου αναφέρθηκε. Φυσικά δεν πρόκειται, δεν είναι θέμα μιας φυλακής, έτσι. Ζούμε σε μια αλληλέγγυα συνδεδεμένη οικονομική κοινωνία. <clears throat> Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα και ελπίζω ότι καταρχήν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για αυτά τα δύο θέματα. Πρώτον λοιπόν και παράλληλα με αυτό που στην λέσχη των 20, G20 αποφασίστηκε και επιβεβαιώθηκε. Κανένας ε, κύριος ε, εμπλεκόμενος πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί χωρίς ε, ρύθμιση να παραμείνει στον τομέα δραστηριότητάς του. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο και για μας από πλευράς νομοθεσίας στην Ευρώπη. Είναι ένας πρώτος ορισμός για την ποιότητα της εργασίας μας. Εμείς συστημικούς κινδύνους θα τους αντιμετωπίζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγούν στο να έχουμε μια παρόμοια κρίση και να την ξαναζήσουμε σαν αυτή που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι συστημικοί ε, κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον θετικό τρόπο και το οφείλουμε αυτό στους πολίτες που μας έστειλαν εδώ σε ευρωβουλευτές. Δεύτερον σημαίνει αυτό ότι δεν οικοδομούμε μια φυλακή, ένα σοφρονιστήριο, αλλά δημιουργούμε προδιαγραφές για την ποιότητα ποιότητα στις εργασίες αυτές και όσοι εμπλέκονται πρέπει να μετρώνται με αυτές τις προδιαγραφές ποιότητας. Και ο συνάδελφος Καμάρ πιστεύω ότι θα συμφωνήσει. Πρόκειται για υψηλή ποιότητα, βέλτιστες πρακτικές και τα υπόλοιπα είναι πραγματιστικό εγχείρημα, ρεαλιστικό εγχείρημα. Δεν είναι θέμα ιδεολογιών. Θέλουμε ρεαλιστικά να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, να αποφύγουμε συστημικούς κινδύνους και από την άλλη πλευρά να έχουμε προδιαγραφές υψηλής ποιότητας στα χρηματοοικονομικά. Αυτό με οδηγεί στις εξής παρατηρήσεις. Εξακολουθώ να το θεωρώ πρόβλημα, πρέπει να πω ότι σε σχέση με τους μάνατζερ, τους ε, επικεφαλείς ε, ε, στην πρόταση της Επιτροπής όπως ρυθμίζεται και δεύτερον υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές προσπάθειες ορισμού των κατοφλίων και πρέπει να δούμε από πιο κοντά αυτά τα θέματα υπό το πρίσμα της καλής υψηλής ποιότητας. Αυτό απαιτεί να έχουμε ένα λειτουργικό level playing field, ένα ισότιμο δίκαιο πεδίο δραστηριοποίησης. Αυτό δεν επιτρέπεται να παρακολύεται επειδή έχουμε κάποιες ε, προδιαγραφές ε, για την ποιότητα που θα μας κάνουν να δεχόμαστε πιο χαμηλές εξωτερικές προδιαγραφές ή σε σχέση με κάποιους μάνατζερ να επιτρέπεται σε κάποιους με χαμηλότερες προδιαγραφές να δρουν. Εδώ πρέπει πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των καταναλωτών να διασφαλίζεται διότι είτε θα πρόκειται για ε, αλήθεια που θα αναφέρεται ότι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας θα πρέπει να ισχύει και να τηρείται και εδώ το πρόβλημα στη ρύθμιση εξωτερικά εσωτερικά πρέπει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Και αυτό αφορά και το τρίτο θέμα δραστήρια ή παθητική ε, δράση marketing. Αν δεν θέλουμε να παραπλανήσουμε κανένα, πρέπει εδώ και η παθητική δραστηριότητα marketing να ε, εξετάζεται. Window dressing στα αγγλικά. Δεν πρέπει να υπάρχει ρύθμιση που θα ε, είναι ρύθμιση για τη βιτρίνα, για ρεκλάμα, αλλά που δεν θα αλλάζει τίποτα ποιοτικά επί της ουσίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πέμπτον μια καλή αξιολόγηση κινδύνων των δραστηριοτήτων. Αυτό αφορά και την μοχλική επίπτωση, επίδραση και τα ίδια κεφάλαια και τις ρυθμίσεις για τους μάνατζερ. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Και εν τέλει δεν είναι αποδεκτό πρέπει να πω αν οι υποχρεώσεις πληροφόρησης έναντι των εποπτικών αρχών δεν ρυθμίζονται όπως πρέπει σωστά. Και αυτό είναι ένα σημείο που το θεωρούμε σημαντικό σκηνοβουλευτική ομάδα όταν one size fits all έχουμε ένα πρόβλημα δηλαδή σε σχέση με μια ρύθμιση για όλους ισοπεδωτικά δεν είναι δυνατόν ισοπεδωτικά να τα αντιμετωπίζουμε όλα όμως πραγματιστικά και ρεαλιστικά είμαστε ανοιχτοί να δούμε την πιο σκόπιμη και καλή ρύθμιση που πρέπει να πετύχουμε γιατί αυτό θα καθορίσει τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, next Σας ευχαριστώ. Πίτερ Σκίνερ επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σε σχέση με την προσπάθεια καθορισμού αυτού του πλαισίου. Jean σου έχουμε εμπιστοσύνη να καταλήξει σε μια ισορροπημένη πρόταση. Φυσικά θα προσπαθήσουμε από κοινού μαζί σου να καλύψουμε τα κενά, αλλά να είμαστε σαφείς. Κάποια από τα κέντρα βάρους που πρέπει να καθοριστούν ήδη τα καθόρισες. Το θέμα για παράδειγμα των ε, κεφαλαίων και των ρυθμίσεων είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα onshore στην Ευρώπη για να μην πούμε τίποτα για το offshore σε σχέση με το πώς τα κεφάλαια διαχειρίζονται και πώς ρυθμίζονται. Και αυτό το θέμα των, του private equity και των hedge funds πρέπει να μας κάνει να το ξαναδούμε. Έχουμε 1,6 δις ευρώ όσον αφορά για παράδειγμα το θέμα των καταναλωτών στη Γαλλία που πρέπει να επιληθεί. Το Κογκρέσο τον είπα, είπε ότι πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να δώσουμε συνέχεια και εμείς να δούμε πώς θέλουμε να επικεντρωθούμε επικεντρωθούμε σε μια συνεπή προσέγγιση, συνεκτική προσέγγιση για τη ρύθμιση αυτού του τομέα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε μια συνέπεια και συνεκτικότητα για να προχωρήσουμε. Δεν φτάνει να θέσει η Ευρώπη τα του οίκου τη εντάξει, αλλά και άλλε χώρε πρέπει να προστεθούν στην Ευρώπη. Το θέμα των τρίτων χωρών είναι σημαντικό. Και να μην αφήσουμε το γεγονό των νέων κλάστερ, των νέων ομάδων που εμφανίζονται offshore και το πώ θα διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια. Και το το θέμα των διαχειριστών, να δούμε σε σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές τι θα γίνει. Πρέπει να επιμερίσουμε το έργο καλύτερα, να καθορίσουμε και να προσδιορίσουμε τα πράγματα καλύτερα. Το υπενήχθηκε αυτό, το σκιαγράφησες όταν είπες για το πώς θα θέλουμε να προχωρήσουμε. Και το θέμα της αναλογικότητας, αναλογικότητας Βουλφ, και το θέμα για την φερεγγιότητα 2, το είχαμε συζητήσει για τα κατόφλια. Δεν μπορέσαμε να καθορίσουμε όμως, να προσδιορίσουμε την αναλογικότητα, δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε ένα σωστό ορισμό για την αναλογικότητα. Πρέπει με φύη, εφάνταστο τρόπο να μπορέσουμε να βρούμε κάτι, αν όχι να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω, να περιμένουμε δηλαδή λίγο περισσότερο να οριμάσουν τα πράγματα και να δούμε για άλλε οδηγίε σε άλλου τομεί πώ μπορούν να προσαρμοστούν όλα αυτά. Για τη συζήτηση α μην είμαστε λοιπόν ανόητοι και παγιδευτούμε σε μια ε, πολεμική αντιπαράθεση ε, αμφίβολη σημασία για το τι μπορεί να επιτευχθεί. Δεν προσπαθώ να διαφωνήσω εδώ μαζί σου, αλλά έχει νόημα να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς στην προσέγγιση μας. Venture capital τώρα, κεφάλαια κινδύνου να πω ε, εδώ δύο λόγια για το risk, risk capital. Είναι κάτι το οποίο είτε ε, έμεσα είτε άμεσα μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Διερωτώ με αν κάποια από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν κεφάλαια για αυτά τα κεφάλαια κινδύνου, αν θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να συμπεριληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προκαλέσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το φάσμα, για το πεδίο εφαρμογής, να δούμε τι μπορεί να γίνει και για τις επιπτώσεις που πάγονται όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετοί ομιλητέ ε, το ανέφεραν. Χρήσιμο θα ήταν να σκεφτούμε και να δούμε αν είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, δούμε, να δει το θέμα το ότι μία ρύθμιση μπορεί να μην καλύπτει όλου. One size doesn't fit all, λέει ο μιλητή. Να μην τα αντιμετωπίσουν αυτά ισοπεδωτικά δηλαδή και να δούμε την δυνατότητα διαφοροποίηση ε, και να υπάρξει η δυνατότητα να διαμορφωθούν ρυθμίσει για, αυτό, για αυτή την κινητήρια δύναμη. Θα δούμε δούμε τις λεπτομέρειες λοιπόν. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Φυσικά οι απόψεις πολλές φορές ε, διαφέρουν. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιες παροχημένες ε, απόψεις ή τέλος πάντων ε, να μην, είναι, να μην μπλέκονται τα πράγματα όταν θέλουμε να τα συζητήσουμε για μια ρύθμιση σαφή και σκόπιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πίτερ Σκίνερ. Επόμενος η Ντανούτα Γεσβέσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ο ρόλος των ε, διαχειριστών ε, θα είναι οπωσδήποτε πολύ πιο καθορισμένος όσον αφορά τώρα τις διαφορετικές συναλλακτικές ε, επενδύσεις και θα είναι διαφορετικός τουλάχιστον από αυτό που είχαμε προβλέψει για τα CSD. Η οδηγία αυτή ε, προτείνει νέες υποχρεώσεις για κάποιους διαχειριστές, αλλά αυτό δεν προεβλέπεται ε, εις το ε, αρχικό κείμενο για τα CDS. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κυρίως την αξιολόγηση των κεφαλαίων κινδύνου και επίσης μας λένε ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο των ορισμών και των, και των ε, θέσεων. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ και με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν εδώ στοιχεία τα οποία καλό είναι να παραμείνουν και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την συναπόφαση και την επιτροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Δανούτα. Η Κάθριν Στήλα έχει το λόγο. Thank you, um, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στάιλερ, όχι Στήλερ. Παρακαλώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ε, και το, τους προλαλήσαντες. Βεβαίως, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα ε, το οποίο δεν έχει θυχτεί. Investment Trust Companies είναι ένα θέμα ε, το οποίο ε, καμιά φορά μπερδεύεται ο κόσμος, ε, ίσως και η μετάφραση να φταίει και το μπερδεύουν με τις investment banks, με τις τράπεζες επενδύσεων. Μιλάω για investment trust companies. Υπάρχουν ε, ας πούμε στην Σκοτία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ε, και ε, νομίζω ότι μιλώντας, συζητώντας για την οδηγία αυτή να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και να μην ξεχνάμε θεσμούς που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια και που σαφώς δεν αντιτίθενται στις αρχές της ε, χρηστής και καλής διακυβέρνησης ε, αυτές ε, οι επιχειρήσεις τις οποίες αναφέρομαι εγώ έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς, έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σύστημα εποπτείας και επιθεώρησης ε, και επομένως να προσπαθήσουμε να μην πετάξουμε και το μωρό μαζί με το νερό που του κάναμε μπάνιο και να είμαστε προσεκτικοί να αποφύγουμε και οποιονδήποτε συστημικό κίνδυνο όταν υπάρχουν πρότυπα καλής διαχείρισης να τα διατηρήσουμε. Επομένως λοιπόν, έστω και αν πιστεύω όντως ε, ότι ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, και ακόμα και αν συμφωνώ με αυτά που είπε προηγουμένως ο Πίτερ Σκίνερ, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές οι investment trust companies είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο είδος το οποίο έχει πολύ καλές πρακτικές. Ευχαριστώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα ή μετά. Μόλις έφτασα, επομένως, ε, θα ήθελα να έχω λίγο το χρόνο να ακούσω πριν, ε, πριν ε, δώσω την, το τελευταίο μου λόγο. Ναι, ναι, απλώς σας ρώτησα, απλώς είδα ότι, ότι φτάσατε, είστε σκιώδης συγητής Ε, ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούσε κανείς να καθορίσει το πότε θα έρθει στην αίθουσα γιατί ήταν ενδεικτική μάλλον η ημερήσια διάταξή μας. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω εδώ Πρόεδρε ότι την Άνοιξη αυτό που σκοπεύω είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και είδαμε τα προβλήματα που υφίστανται, μπόρεσα να εξοικειωθώ κάπως περισσότερο με το θέμα και τη συζήτηση που κάναμε ανάλογα να την προσανατολίσουμε. Υπάρχει φυσικά κάποια πολιτική πίεση. Η Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη θέλουν σχετικά γοργά να υπάρξει μια ρύθμιση. Μια ρύθμιση ώστε τέτοιο είδους κίνδυνοι να μην επαναληφθούν όπως αυτή της κρίσης και όσον αφορά την οικονομική κατάσταση στην οποία καταλήξαμε, την οποία και προκάλεσε αυτή η κρίση, να μην επαναληφθούν όλα αυτά. Κατά τα άλλα, με τις εθνικές ρυθμίσεις ε, ασχολήθηκα περισσότερο και τώρα με εκπλήσει κάπως ότι όλα θέλουν τόσο γοργά να τα ε, καταφέρουμε και να τα ολοκληρώσουμε. Με υπερβολική βιασύνη θα έλεγα. Καλύτερο θα ήταν να τα δούμε περισσότερο σε βάθος, πιο προσεκτικά, προτού βιαστούμε υπερβολικά. Θα ήθελα σε σχέση με τις παρατηρήσεις των συναδέφων, συναδέφου καμάλ και άλλων που ε, τοποθετήθηκαν σχετικά να πω μόνο τα, τα εξή εν συντομία. Ο βαθμός προστατευτισμού σε αυτό το έγγραφο είναι θα έλεγα ιδεολογικού χαρακτήρα. Έχει ένα, έχουμε ένα είδος προστατευτισμού που δεν γνωρίζαμε στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Με εκπλήσει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάποια τέτοια πράγματα Πιστεύει κανείς άραγε ότι αυτός ο προστατευτισμός σε αυτό το έγγραφο όπως περιγράφεται θα δώσει κάποια πλεονεκτήματα για αυτή την Ευρώπη. Σίγουρα όχι. Και εξάλλου όχι μόνο για το ότι κάποιοι φαντάστηκαν να προτείνουν τέτοια πράγματα. Αυτό είναι όμως το αποτέλεσμα όταν καταλήγουμε σε υπερβολική βιασύνη και θέλουμε υπερβολικά βιαστικά να ρυθμίσουμε τέτοια πράγματα. Αλλά είναι και χρωματισμένο ιδεολογικά αυτό το θέμα για αυτόν τον προστατευτισμό. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά στο τέλος. Οι επενδυτές, έτσι. Διότι αυτό περί το οποίο πρόκειται είναι εδώ σε σχέση με την Αφρική ε, και τους, ε, τα θέματα και των ε, δικών μας πολιτών και της, το, της συνταξιοδότησης δεν μπορούν όλα αυτά να ταιριάξουν σε, ένα, σε μια προσέγγιση ισοπεδωτική one size fits all με ένα μέτρο το οποίο θα ρυθμίζει τα πάντα. Δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδικοί, ισοπεδωτικοί. Υπάρχουν διαφορετικά θέματα εδώ και δεν είναι δυνατόν να τα αμελήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τι η πορεία θα οδηγούσε εξάλλου στο τέλος στο να, με την οδηγία αυτή μάλλον οι κίνδυνοι να αυξηθούν ή να πολυμορφοποιηθούν και να μην αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους. Και αυτό είναι ένας επιπλέον κίνδυνος όταν βιάζεται κανείς υπερβολικά και δρά χωρίς να τα έχει ε, μελετήσει όλα όρημα. Και σε σχέση με την ε, ρύθμιση και βελτιώσεις στην αγορά, δεν θα είναι βελτιώσεις πιστεύω αυτές, γιατί θα οδηγήσουν τελικά στο τέλος τέλος να υπάρξει μια αναταραχή σε σχέση με τα όσα θα συμβούν μετά την οικονομική κρίση μάλλον αναταράξεις θα υπάρξουν αντί να βελτιωθούν τα πράγματα σε σχέση με την αγορά. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγούσε σε βελτιώσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και κάτι άλλο σε όλους, ότι με αυτούς, με αυτούς τους περιορισμούς που ε, προσεγγίζονται με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ρύθμιση που εκείνοι που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση να πληρώσουν για τις ζημιές και να, να είναι υπεύθυνοι, διότι δεν είναι δυνατόν άλλοι να υπομισθούν τα σπασμένα. Πολλά πρέπει να γίνουν λοιπόν ακόμα για να υπάρξουν οι σωστές βελτιώσεις που είναι αναγκαίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση από πλευρά του εισηγητού του αξιόλογου εγγράφου είναι μια καλή αφετηρία. Δύο πράγματα θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ. Είναι δύο ελλείψεις, δύο ε, κενά που υπάρχουν, που πιστεύω εγώ ότι στο έγγραφο εδώ λείπουν δύο στοιχεία. Θα έπρεπε όμως με αυτά να ασχοληθούμε και να τα δούμε. Αφενός πρόκειται πρώτα για τους διαφορετικούς τύπους ε, ή την τυπολογία που δεν, περιγράφονται επαρκώς στην ε, οδηγία αναφέρονται ως ε, μη κοινή χρήση. Έτσι οι διατάξεις για τον ανταγωνισμό δεν προσαρμόζονται σχετικά και αυτό οδηγεί στο ότι κάποια κράτη-μέλη να ε, πλήττονται ιδιαίτερα μειονεκτικά κιόλα, να είναι σε αρνητική θέση. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν αυστηρές ρυθμίσεις και εκεί κάποιες επιχειρήσεις που περιοριστικά θα αντιμετωπίζονται θα μετεγκατασταθούν και θα αναζητήσουν έδρες σε χώρες όπου δεν θα είναι εξίσου περιοριστικές οι διατάξεις και οι όροι. Θέλουμε λοιπόν διατάξεις και όρους που θα είναι κοινοί για όλους ε, ώστε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Και δεύτερον, όσον αφορά κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να καλύψουμε που απουσιάζει, θα έλεγα σχετικά με αυτό ότι αυτή η οδηγία δεν ε, παρακολεί ένα εναλλακτικό ταμείο σε σχέση με την, ε, τις επενδυτικές δραστηριότητες ε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να παρακάμπτουν κάποιοι τις διατάξεις που θα ισχύουν. Και αυτό πάλι θα οδηγήσει στο ότι οι ιδιωτικοί, οι επενδυτές ε, και οι πολίτες να επομίζονται κινδύνους που είναι υπερβολικοί. Τέτοιους κινδύνους πρέπει να τους αποφύγουμε θα έλεγα και να τους απομακρύνουμε από το, το σύστημα μας, να τους εξαλείψουμε. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το εξαίρετο έγγραφο εργασίας. Το διάβασα προσεκτικά, αλλά δυστυχώς έφτασα αργοπορημένη και δεν άκουσα αυτά που είπε στην αρχή. Εν πάση περιπτώσει, εκπλήσωμαι από το εξής κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ε, καθυστερεί λίγο πριν κάνει τέτοιου είδους προτάσεις αλλά τώρα φαίνεται να έχει ε, ε, φαίνεται ότι έχει επιταχύνει ιδιαιτέρως βεβαίως η οδηγία αυτή είναι πολύ σημαντική και εγώ έχω κάποιες επικρίσεις τις οποίες θέλω να διατυπώσω αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε όλοι μια επικοδομητική πρόταση έτσι ώστε να βελτιωθεί πραγματικά η οδηγία αυτή γιατί για μένα υπάρχει μια αρχή η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική ε, και τις οποίας πρέπει να υπεραμεινθούμε. Εάν υπάρχει λοιπόν νομοθεσία για τα hedge funds θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να διευρυνθεί έτσι ώστε και να προστατεύεται ο κόσμος από τα hedge funds αλλά και ε, από άλλου είδους επενδύσεις και βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε και στο μέλλον τέτοιου είδους συστημικούς κινδύνους και τέτοια επικίνδυνα προϊόντα. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να έχω και περισσότερες πληροφορίες ε, εάν ε, κάνουμε, προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές ε, ή προσαρμογές. Δηλαδή θέλω να ξέρω ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των αποφάσεών μας. Ε, αναφέρεται ότι τα εθνικά, ε, εθνικοί πόροι θα πρέπει να τα εθνικά φαντς μάλλον θα πρέπει να αποκλείονται. Ε, ναι, αλλά εγώ θέλω να έχω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει όλη αυτή η αναμόχλευση. Άλλο στοιχείο, ε, τα, οι τρίτες χώρες και άλλωστε αναφέρθηκε ε, και από τον ίδιο τον εισηγητή στο έγγραφο εργασία που έχουμε. Θέλω να ξέρω λοιπόν τι θα γίνει με τις τρίτες χώρες, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα συμβεί ε, εάν περιορίσουμε ε, τις ε, διαδικασίες μονάχα στις επενδύσεις και τους επενδυτές που έχουν την έδρα τους σε τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, ορθώς στο έγγραφο εργασίας γίνεται λόγος και για άλλα καθεστώτα, ούτσις, τα κτλ. Πώς, πώς είναι δυνατόν να είμαστε λογικοί λοιπόν και συνεκτικοί ε, με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο. Εγώ θα προχωρήσω δε ακόμα περισσότερο και θα πω ότι ε, τη στιγμή που ε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία. Τι θα γίνει δηλαδή, αυτοί θα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή, θα πρέπει να χάσουν όλο το χρόνο που έχουν ήδη αφιερώσει. νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν άλλα κριτήρια. Τώρα ένα άλλο σχόλιο το οποίο αφορά σειρά ε, την, ε, τις νέες υποχρεώσεις που θέλουμε να ε, εφαρμόσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η αρχή της αναλογικότητας. Θα πρέπει να δούμε βεβαίω και αν η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που θέσαμε, αν μπορεί να αντιδράσει και με ποιο τρόπο θα αντιδράσει. Κάτι άλλο σημαντικό. Διάβασα στην εφημερίδα ότι η Σουηδική Προεδρία προτίθεται να υποβάλει σημαντικές τροπολογίες ε, στην ε, πρόταση αυτή, στην πρόταση οδηγία. Ε, και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που προτίθεται ε, να προτείνει η Σουηδική ε, Προεδρία. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα ανταποκριθούμε και εμείς στα σχόλια αυτά. Ευχαριστώ. Άλεν Μακάρθη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ και εγώ δεν άκουσα τι είπε ε, στην αρχική του εισήγηση ο κύριος Γκοζέ. Ε, εν πάση περιπτώσει πάντω πιστεύω, πιστεύω λέω, ε, ναι, δεν είπα και τίποτα σημαντικό, λέει ο κύριο Γκοζέ. Ήταν πάρα πολύ σύντομη, δεν χάσατε και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία από τον οποίο όλοι συμφωνούμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για εναλλακτικέ επενδύσεις ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι λίγο μια διαφορετική μορφή ε, εργασίας και βεβαίω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, διακανονιστούν με κάποιο τρόπο τα, τα κεφάλαια αυτά έστω και αν προκάλεσαν κατά κάποιο τρόπο ή ήταν μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, τη θύελα τη κρίση, χωρίς να καταργηθούν θα πρέπει οπωσδήποτε οπωσδήποτε να τα ρυθμίσουμε καλύτερα. Ε, νομίζω ότι οι διαχειριστές ε, των ε, hedge managers, των hedge funds, ήταν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης πριν από αρκετά χρόνια. και νομίζω ότι τώρα μάθαμε το μάθημά μας. Πρέπει να είμαστε proactive. Πρέπει πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να τους πιέσουμε έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά τους σωστά με τρόπο αξιόπιστο. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με θέματα αυτά και από την προηγούμενη επιτροπή μου έχουμε δουλέψει επίσης σε τριμερή διάλογο, ε, σε προσπάθεια επίτευξης κάποιας ε, συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την, ε, τον κανονισμό αυτό. Όχι γιατί δεν θέλω να, υπάρχουν, να υπάρξει διακανονισμός των private equities και των hedge funds και των οποιονδήποτε άλλων άλλων προϊόντων. Λέω απλώς ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτών των ε, προϊόντων γιατί μπορούν να ε, δώσουν όθηση στην οικονομία όταν λειτουργούν σωστά. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και να διαβάσουμε προσεκτικά και την ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης να δούμε και ποιε θα είναι οι επιπτώσεις στου επενδυτές οποιονδήποτε τροποποιήσεων επιφέρομαι στο υπάρχον σύστημα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει μέσω των αποφάσεών μας να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις απειλές και τους κινδύνους που μελλοντικά θα απειλήσουν το ε, οικονομικό ε, σύστημα. και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο τις διατάξεις οι οποίες αφορούν ακριβώς αυτή την έδρα στην ε, Ευρώπη γιατί διαφορετικά θα πρέπει να αλλάξουν και οι εθνικές νομοθεσίες ε, και, ε, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε και τον εθνικό νομοθέτη από τον οποιοδήποτε διακανονισμό γιατί αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα πώ έχει η αγορά του, αν υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητε, αν υπάρχουν οι λεγόμενες έκτακτες συνθήκες κτλ και νομίζω ότι δεν είναι καλή ιδέα να είμαστε απόλυτοι ε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε και από αυτούς. Ε, βλέπω ότι ο ε, εισηγητής έχει ασχοληθεί ε, με την σχέση που θα πρέπει να έχουν οι Εθνικές Ευρωπαϊκές Αρχές και την, με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Συστημικών Κινδύνων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό είναι να υπάρξουν υποχρεώσεις, αλλά οι υποχρεώσεις αυτές να μπουν σε ένα ισορροπημένο σύστημα όπου θα έχουμε ε, θα έχουμε ε, ελέγξει εκ των προτέρων τον αντίκτυπο γιατί δεν έχει έννοια να επιβάλλει κανείς πάρα πολύ ε, βαριές υποχρεώσεις χωρίς να έχει εντωμεταξύ προβλέψει τον αντίκτυπο στις αγορές. Χαίρομαι επίσης γιατί ο κύριος Γκοζές προσπάθησε να διασυνδέσει την οδηγία αυτή με άλλες υφιστάμενες οδηγίες και νομίζω ότι Καλό είναι να βλέπουμε ποια είναι η διάδραση ανάμεσα ε, στο σύστημα αυτό, γιατί όλες αυτές οι οδηγίε θα πρέπει και οι κανονισμοί θα πρέπει να δουλέψουν σαν ένα σύστημα. Και μία ακόμα φορά θα πω ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που, ε, ανέλαβαν ε, η Πρόεδρος με τον εισηγητή για την εκπόνηση δηλαδή μελέτης επιπτώσεων και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα γιατί διαφορετικά όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η μείωση των συστημικών κινδύνων εάν δεν γίνει η σωστή πρόβλεψη μπορεί να στραφεί εναντίον μας. Thank you. Next on, my list. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκαρθία επόμενος ομιλητής. Όμως, σας λέω εκ των προτέρων, ότι μόλις αυτή η ζήτηση τελειώσει, πριν ε, οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να μιλήσει και το Συμβούλιο. Και μετά ε, η συγητής, η Κομισιόν και πάλι, συγγνώμη, πρόεδρε που και εγώ μια που επιταχύναμε τις εργασίες μας, δεν άκουσα το, την σύγχυση του κυρίου Γκοζές που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ αξιολογική τώρα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις γενικού χαρακτήρα. Ξέρω ότι πρέπει να διευρυνθεί η ελεγκτική ρυθμιστική μας λειτουργία για όλους όσοι μέχρι τώρα κινούνται σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο. Θα πρέπει αυτό να γίνει ταχαίως, να μην χάνουμε χρόνο. Γιατί το θέμα είναι δύσκολο. Τρίτον, επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κριτήριο σύγκλησης όσον αφορά κάποιους τομείς που είναι σημαντικοί για την ανταγωνιστικότητά μας όσον αφορά την ΟΝΕ. Συμφωνώ με την τελική έκθεση της ε, οδηγίας, όμως συγκεκριμένα δεν συμφωνώ με τα όσα αναφέρονται όσον αφορά τη ρυθμιστική λειτουργία. Λέει η τελική έκθεση ότι τα εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων είναι ε, κάτι το γενικό που καλύπτει ένα σωρό διαφορετικά είδη. Όμως η νομοθεσία ισχύει έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα επένδυσης και άρα προσοχή να μην αναγκατεύουμε πράγματα που δεν πρέπει και το αντίστροφο να διαφοροποιούμε κάποια που δεν θα έπρεπε. Οπότε, προσοχή για κάποια ταμεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία αναφέρονται στην τολική έκθεση γιατί υπάρχουν κάποια τέτοια ταμεία ενώ όπως ας πούμε τα, τα κεφάλαια επενδύσεων γιατί μιλούμε για κάποια ταμεία πρώτων υλών ε, που ε, διατρέχουν κάποιους κινδύνους και λέει εδώ πέρα ότι είναι ακριβώς όπως τα επενδυτικά κεφάλαια. Όμως η νομοθεσία που αφορά τα ελεύθερα ταμεία και τα των πρώτων ε, υλών είναι κάτι το οποίο καλύπτει και για τα κατόφλια και για την κάλυψη και από άλλες οδηγίες Αναφέρεται επομένω σε όλα τα ταμεία και όσον αφορά τι διατάξει για την διαφάνεια επίση. Εδώ καλύπτονται και τα κεφάλαια επενδύσεων όσον αφορά τις προϋποθέσεις που τάσσονται για ε, κεφάλαιο, για καταθέσεις και για θέση στο χρηματιστήριο. Επίσης, θέλουν να καλύψουν όλα τα ταμεία και όσον αφορά τις διατάξεις για τη διαφάνεια. Το είπαν αυτό διάφοροι ομιλητέ, ότι θα πρέπει με προσοχή να δούμε τι θα ισχύσει και για τα ταμεία των τρίτων χωρών. Να προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε σε σχέση με τα κεφάλαια που υπάρχουν εκτός Ευρώπης. Επίσης, να μελετήσουμε ποιες θα είναι οι μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά κάποια ταμεία που είναι κλειστά όσον αφορά διάφορα χαρακτηριστικά τους. Και, βάση να συντονίσουμε την ιδεολογική έκθεση με το σώμα του νομοθετήματος. θα πρέπει να γίνει η διάκριση όσον αφορά τα ταμεία μεταξύ τους και τους διαφορετικούς κινδύνους που διατρέχουν. Δεν είναι δυνατόν με μία ρύθμιση να τα καλύψουμε όλα, γιατί τα χρηστικά του κάθε οικονομικού φαινομένου είναι διαφορετικά. Ελπίζω να το καταφέρουμε αυτό, να το καταφέρουμε έγκαιρα και να μπορέσει ο κ. Γκοζές ως συνήθως να προτείνει κάποια ρύθμιση ευφυή. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά. Σύμφωνα με την... Ή μάλλον όπως και ο κύριος Μαργάγιο και εγώ δυστυχώς έχασα την εισήγηση του συγητή. Να σας πω πάντως τι πιστεύω για το κείμενο. Εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω μια δεκαετία δουλεύω σε αυτήν την επιτροπή μας και σπάνια έχω δει προτάσεις κομισιών που τόσο πολύ σχετίζονται με τα όσα προσβεύουν τα λόμπι. Υπάρχει καλή πίστη. Σκοπεύουν σε μια προσέγγιση θέσεων, αλλά αλλά, αλλά, αλλά, τόσο πολύ που τελικά αποδυναμώνεται αυτή η πρόταση. Φυσικά και πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την πρόταση σκοπεύει να ρυθμίσει ε, κάποιους ε, οργανισμούς που ο καθένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όσο και αν υπάρχει διαφοροποίηση από τον ένα οργανισμό στον άλλο, θέλουμε να υπάρχει ισότητα, ίση όρια ανταγωνισμού. Άρα δεν, θα είναι, δεν εύκολη η ρύθμιση για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Είχαμε ζητήσει από τον Μακρύβη να μα κάνει κάποιε προτάσει. Εδώ και πολλά χρόνια το ζητάμε και μα έλεγε ο Μακρύβη ότι προτιμάει την αυτορύθμιση. Το έλεγε και το ξανάλεγε. Τώρα προτείνουν αυτό το νομοθέτημα το οποίο ίσως ε, υπερβαλλόντως ρυθμίζει ορισμένους τομείς. Εμείς όμως είμαστε συνομοθέτες. Εμείς και το Συμβούλιο και εμείς θα κρίνουμε τελικά αυτά τα οποία προτείνονται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ε, υπάρχει μεγάλη ενισχύση στην αγορά, αναφέρθηκε από κάποιο συνάδελφο. Εγώ σας λέω ότι ο Κοσμάκης ανησυχεί ακόμη περισσότερο από τις αγορές. Γιατί? Έχουν γίνει μάρτυρες του πού μπορούν να φτάσουν οι συνέπειες για απασχόληση και για εισόδημα της κερδοσκοπίας. Άρα, το πρώτο που πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς τον κοσμάκι αυτόν που δεν καταλαβαίνει αυτούς τους μηχανισμούς της αγοράς, πώς θα τον καλύψουμε. Άρα θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σωστά. Ένα επίσης ανέφερε θα πρέπει να περιοριστούμε στο ποιο θα είναι ο φταίχτη. Δεν καταλαβαίνω τι πάνε να πει οι Ήδη και κάποιον καταδικάσαμε. Όμως, για να καταδικαστεί κάποιος, θα πρέπει να καταδικαστεί με τη βάση κάποιου νόμου, τον οποίο θα έχουμε θεσπίσει. Και κατόπιν να προβούμε εις τις κυρώσεις κατά αυτού που έφταξε. δεν ξέρω, στην αρχή της κρίσης, στις 7 ε, δεκάτου αποφάσισαν κάποια πράγματα οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων. Επιτρέψτε να σας παραπέμψω στο ότι είπαν ότι κανείς χρηματοοικονομικός οργανισμός, ε, κανένα τμήμα της αγοράς και ε, κανένα δίκαιο εθνικό δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στην διαδικασία της εποπτείας. Και όλοι που έχουν κάποια, κάποιο συστημικό ειδικό βάρος, όπως αυτά τα επιχειρηματικά κεφάλαια με το, με το υπομόχλιο θα πρέπει να περνάνε από κάποια εποπτεία όπου και να βρίσκονται. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και λέει παραπέρα. Λένε οι αρχικά των κυβερνήσεων. Η διαφάνεια για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ένα σύστημα πληροφόρησης το οποίο να είναι πληρέστερο. Όσον αφορά την δραστηριότητα αυτών που αναπτύσσουν τέτοια οικονομική δραστηριότητα. Άρα, θα πρέπει πιο προσεκτικά να εξετάσουμε τι γίνεται με αυτό το, το φαινόμενο του υπομόχλειου. Εδώ κάποιος πάρα πολύ σημαντικός ε, ε παράγοντας ε, που είναι διοικητής της Τραπεζάς της Γαλλίας λέει πώς είναι δυνατόν να έχουμε κάποιες συνήθειες από τη σόρευση των συνεπειών του υπομόχλιου όσον αφορά τα derivatives των πιστώσεων. Και ο Χριστιανόγια δίνει ένα παράδειγμα λέγοντας ότι μπορούμε να φανταστούμε ένα τέτοιο ταμείο που έχει ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο 100 δανείζεται 200. Φτάνει επομένω σε κεφάλαιο 300. Το επενδύει σε ένα επενδυτικό οργανισμό που των 300 επίσης δανείζεται άλλα 300 και φτάνει στα 600 επομένως αυτός ο επενδυτικός οργανισμός κατόπιν με αυτά τα 600 γίνεται CDO ε, επένδυση και εκεί έχουμε υπομόχλιο 10 επομένως βλέπετε ότι έφτασε το επίπεδο έκθεσης από το αρχικό κεφάλαιο των 100 έφτασε σε έκθεση του ύψους 6.000, δηλαδή 60 φορές παραπάνω από το κεφάλαιο. Επίσης, λέει εδώ πέρα ο Νοαγέ, ότι φτάνουμε σε μια πυραμίδα χρέωσης. Το 2% επομένως του ενεργητικού είναι, είναι, είναι, ικανό για να κυμηδενήσει το σύνολο του κεφαλαίου. Έτσι, μπορεί να διαπιστώσετε γιατί φτάσαμε σε αυτή την κρίση σε τόσα προβλήματα. Και αυτό το long term management capital, αυτή η, αυτό, τα, τα, τα, τα κεφάλαια μακροπρόθεσμης ε, διαχείρισης μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Διότι είχαν εκτεθεί κατά 180% του κεφαλαίου τους. Βλέπετε επομένως την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος να προσπαθεί να επενδύσει χωρίς να προσπαθεί να βάλει κάποιο φρένο σε αυτό το σύστημα, κάποιο τροχοπέδι. Κύριε Γκέμπρος, ευχαριστούμε, λέει κύριο Γκαρθία Μαρκάγιο. Και τώρα η κυρία έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτω συγγνώμη στον κύριο Γκοζές που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίασή του σήμερα το πρωί. Ήμουνα στην... στον Ποτηλιάρισμα καθώς ερχόμουν από το αεροδρόμιο. Θα ήθελα εδώ τώρα σε σχέση με αυτά για να ζητήσω συγγνώμη αν κάποια... κάποιες παρατηρήσεις έγιναν προηγούμενα. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτίμηση κινδύνου που συμφώνησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, την τελευταία συνεδρία. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να μας ε, δώσει μια ένδειξη πού βρισκόμαστε σε σχέση με την αποτίμηση κινδύνων η διαβούλε, από πλευρά ε, συντάκτη γνωμοδότηση έχει καθοριστεί ποιο θα το αναλάβει και τι, σε ποιο ευρώ θα γίνει αυτό. Και θα ήθελα να κάνω λόγο για το κεφάλαιο κινδύνου και venture και risk capital και όπου ο Πίτερ Σκίνερ προανέφερε αναφερόμενοι σε διάφορες εκθέσεις σε σχέση με αυτό το έγγραφο εδώ είναι επικοδομητικό σε σχέση με την ιστορική αυτή διάσταση για αυτά τα θέματα. Η έκθεση για το κεφάλαιο κινδύνου που ο Πίτερ Σκίνερ ήταν εισηγητής το 2003 έχει τεράστια σημασία ασχολείται με το θέμα ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ μικρό κεφάλαιο κινδύνου στις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις. Και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολο να δοθούν πιστώσεις και δάνεια από τις τράπεζες λέγεται ότι όταν δεν υπάρχουν κίνητρα για τους επενδυτές ε, τον είπα, να επενδύσουν ε, σε τέτοιου είδους δραστηριότητες ε, στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνος. Και θα ήθελα να γνωρίζω σε σχέση με αυτή τη συνιστόσα για το κεφάλαιο κινδύνου μήπως υπάρχει κάποια χωρίς πρόθεση εδώ επίπτωση που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσκομα για τις επιχειρήσεις μας. Επίσης θα ήθελα εδώ και την συνιστόσα του μάρκετινγκ της προώθησης να αναφέρω θα ήθελα να καταχωρηθεί ότι κατά την περίοδο εκτέλεσης εφαρμογής ε, οι διεργασίες αυτές ε, τοποθέτησης θα μπορούν να συνεχιστούν. Τα, τα, τα κονδύλια εκείνα τα οποία θα πρέπει να αναγνωριστούν από άλλες χώρες ε, ακόμα για παράδειγμα από τη ΣΥΠΑ μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται υπό την, το πλαίσιο αυτής της οδηγίας για την αγορά. Έγινε λόγος για την μοχλική επίπτωση leverage και δημιουργείται κάποια σύγχυση. Υπάρχουν πάμπολοι ορισμοί που διακινούνται. Θα ήθελα και εδώ να υποβάλω μια πρόταση σχετικά και να πω ότι η μοχλική επίπτωση από πλευρά των hedge funds προέρχεται από μια πηγή ε, πίστοσης. Δεν χρησιμοποιούν ε, ίδιες πιστώσεις ε, για αυτή τη μοχλική επίπτωση. Υπό το πλαίσιο αυτής της οδηγίας λοιπόν ήδη έχουμε την δυνατότητα να εποπτεύουμε και να ελέγχουμε την μοχλική επίπτωση από πλευράς αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γίνεται λόγος εδώ, κάνουν χρήση του ε, brokerage. Αν έχουμε λοιπόν ε, έναν broker που ε, εμπλέκεται, μπορούμε μέσα στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων να ελέγξουμε τη μοχλική επίπτωση θα έλεγα λοιπόν ίσως ε, εξειδικευμένα αναφερόμαστε στο θέμα της μοχλικής επίπτωσης, ε, αλλά μπορούμε αυτό να το δούμε και σε διαφορετικό πλαίσιο. Επίσης θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο ήδη είχα αναφέρει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να είναι ισοδίκαιο το πεδίο δραστηριότητας στο τέλος τέλος. Και εδώ σε σχέση με τα ε, κεφάλαια και τις ε, ε, προδιαγραφές για τα equities μπορεί να υπάρχουν διαφορές ιδιαίτερα όσον αφορά τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Πολλές από τις ευρωπαϊκές τράπεζες εργάζονται με τα κεφάλαια κινδύνου και με τα equity funds και σε σχέση με την απεικόνηση στους απολογισμούς τους δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μεν και δε. Πρέπει να έχουμε ένα ασφαλή ασφαλέ και δίκαιο πεδίο δραστηριοτήτων για όλους όσου εμπλέκονται υπό το πρίσμα αυτό. Και μια τελική παρατήρηση εδώ. Οι μη στοχευμένε ε, μη εσκεμμένε ε, επιπτώσεις ε, που πολλέ φορέ υπάρχουν έχουμε μια ανεξάρτητη εταιρεία που διαχειρίζεται τα διαθετικά κονδύλια που προσέχονται στη δική μου περιφέρεια. Τους ε, τελευταίους μήνες είχαν και τη διαχείριση του Ταμείου Τζέρεμι, τις ε, κοινές ευρωπαϊκές, τα κοινά ευρωπαϊκά κονδύλια για τις ε, μικρές επιχειρήσεις. Μου γνωστοποίησαν ότι σε σχέση με μια γνωμοδότηση υπό αυτό το πρίσμα αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο που θα δημιουργήσει τεράστιες δαπάνες. Και στο τέλος τέλος για τα κονδύλια αυτά τα οποία θα επενδύονται θα υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στο εύρος των ρυθμίσεων που υιοθετούμε ώστε να μην είμαστε υπερβολικοί σε σχέση με τους συστημικούς κινδύνους προβλέποντας το τι θα συμβεί όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Ευχαριστώ. Όλε μη το επόμενος. Παρακαλώ όλε. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπούμε καθυστέρησε η πτήση μου και δεν κατάφερα να παρακολουθήσω τις παρατηρήσεις του κυρίου Γκοζές. Το έκανα όμως το προηγούμενο ε, απόγευμα και έτσι γνωρίζω μπορώ να πω εν μέρη κάποια από τα πράγματα που ανέφερε. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς σε Γενοβουλευτική Επιτροπή ε, είσαι ο, ακριβώς ο ιδανικός, ε, το ιδανικό μέλος, είσαι ρεαλιστής και το, όσον αφορά το εύρος της Επιτροπής στη δράση της νομίζω ρυθμίζεται σωστότερα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και κάποιο θα μπορούσε να πει ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό να έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη μορφή οικονομία. Όμω εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι ήταν τεράστια επιτυχία φυσικά αν δει κανεί το τι συνέβη παγκόσμια στον κόσμο. Και αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, ρυθμίσει ε, και διαφορετικοί τύποι χρηματοοικονομικών μέσων, είναι μέρο τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Κάποιοι ίσω θα έλεγαν δεν θα, θα είμαστε σε καλύτερη θέση αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδου επιχειρήματα. Χρειαζόμαστε ρυθμίσει Δεν θα είναι έκπληξη για σας ίσως το ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ενθερμός οπαδός ε, ρυθμιστικών διατάξεων και περιορισμών. Δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο υπερενεργητικοί. Τώρα, σε σχέση με την ε, ε, υποβολή σχετικών προτάσεων, θα έλεγα ότι ίσως ήταν και μια πολιτική όχληση, political harassment αυτό το οποίο συνέβη Εν πάση περιπτώσει, φίλοι, ίσως καταφέραμε και πήραμε αυτό το οποίο ε, ζητούσαμε, διότι πιέζατε τόσο πολύ και στην αρχή όταν το χρειαζόμαστε. Ήρθε κάποιες ε, μέρες ε, πριν, πριν από τις εκλογές και ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αυτή η ρύθμιση όπως είπε ο κύριος Γκέμπες. Θα έλεγα σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή είμαστε υπεύθυνοι για την διασφάλιση καλύτερου νομοθετικού έργου, καλύτερης νομοθεσίας. Όταν εγώ ήμουν υπεύθυνο για το USIS 2 και το USIS 3 ε, ε, και μετά είχαμε στη συνέχεια το USIS 4, είχαμε διαρκή διάλογο με τις ε, επιχειρήσεις. Ίσως κάποιοι μπορούν να πούν ότι είναι πραγμα... Εγώ δεν είμαι. Προσπαθώ να μάθω περισσότερα πράγματα, να εξοικειωθώ με τα επιχειρήματα σε εθνικό επίπεδο και τα επιχειρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Αγαπητέ κύριε Γκέμπερς, φίλε και συνάδελφε, είναι πολύ καλό το ότι έχουμε εδώ συσσόρευση τέτοιων εγγράφων. Πρέπει να είναι ανοιχτό αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να είναι ε, ανοιχτές αυτές οι εκδηλώσεις ε, και ανοιχτού χαρακτήρα για τα διαφορετικά επιχειρήματα. Και στο τέλος ίσως καταφέρουμε να έχουμε μια βελτιωμένη νομοθεσία και πραγματικά πιστεύω ότι το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω δεν υπήρξε επαρκή χρόνο. δεν ξέρω τι συνέβη. Εμεί πρέπει όμω να καλύψουμε αυτή την ανάγκη έγκαιρα. Είναι ζωτική σημασία να το καταφέρουμε. Και βασίζομαι στον κύριο Γκοζέ και στου υπόλοιπου κοιόδης εισηγητές ότι θα συμπεριλάβατε και εμά και του υπόλοιπου μέσα σε αυτό το έργο όπως και για τα θέματα ε, προβλημάτων φερεγγιότητας για τις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την νομοθεσία να τα καταφέρουμε έτσι. Αρκετά επιχειρήματα θα μπορούσα να σας δώσω από τη χώρα μου, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα τα προσέχατε, οπότε δεν θα το κάνω. Λοιπόν, πραγματικά ελπίζω, είναι μια πραγματική έκκληση σε όλους σας και το χρωστάμε αυτό θα έλεγα και στους πολίτες μας, στην κοινωνία μας, στις επιχειρήσεις, ε, στους, ε, ε, στις εταιρείες που εμπλέκονται σε όλους όσους εξατώνται από αυτές τις ρυθμίσεις. Θα έλεγα λοιπόν Πρόεδρε, για αυτό το χρονοδιάγραμμα, έχω κάποιες ανησυχίες για αυτό το χρονοδιάγραμμα. Φυσικά δημοκρατικά θέματα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και λειτουργικά και να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα. Αλλά αυτή οι τριμερείς διάλογοι τώρα, εγώ δεν είμαι υπέρα αυτών των τριμερών διαλόγων. Είναι ένα είδους ανομαλία αυτό που προκαλείται έτσι. Θα νόμιζα ότι με τη δεύτερη ανάγνωση η νομοθεσία είναι βαίνει καλός. Τόσο αρνητικό είναι αυτό. Είναι πολύ πιο ανοιχτή θα έλεγα. Δίνει ένα περιθώριο, δίνει κάποιους επιπλέον μήνες. Έτσι δεν είναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι το να πιστεύει κανείς ότι αν τα βιάσει όλα και βιαστικά τα ρυθμίσει είναι όλα καλύτερα και ότι θα είναι πιο ευτυχισμένοι οι πολίτες δεν είναι, είναι κάτι αποδεκτό. Τουλάχιστον όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές, έχουν γίνει ευρωεκλογές και έχουμε μια νέα Ευρωβουλή και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλή νομοθεσία αντί να προσπαθούμε όλα βιαστικά να τα καλύψουμε και εν τέλει κύριε Γκοζές, ε, βασίζομαι σε εσά κύριε Γκοζές. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να ακούσετε τα επιχειρήματα, ακόμα και κάποια επιχειρήματα μιας μικρής χώρας από τις σκανδιναβικές χώρες. Έχουμε ε, ε σχετικές ε, ρυθμίσεις και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με τα equity είμαστε υπό δημοκρατικό πνεύμα σοσιαλδημοκρατών, ακόμα και από πλευρά σοσιαδημοκρατίας κάποιοι πιστεύουν ότι χρειάζεται αυτό το ανοιχτό πνεύμα για τη ρύθμιση των διαφορετικών χρηματοοικονομικών μέσων για να προσφέρουμε κεφάλαια στην Ευρώπη δεν πρέπει να παρακολύεται η αγορά από τις ρυθμίσεις μας. Χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια και δεν χρειαζόμαστε προστατευτισμό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτού χαρακτήρα οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Φόρντ παρακαλώ. Thank you very much. And again... Σας ευχαριστώ και πάλι. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Συγγνώμη για το ότι δεν ήμουν παρούσα όταν ξεκίνησε η συζήτηση σήμερα το πρωί δεν ήμουν παρούσα έγκαιρα. Υπήρχαν σημαντικέ καθυστερήσει στο αεροδρόμιο των Βρυξελών σήμερα το πρωί. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια τεράστια σημασία συζήτηση και θα θέλαμε να είμαστε εδώ παρόντε έγκαιρα. Πρόεδρε, με ευχαριστείτε ότι δώσατε πρόσθετο χρόνο να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Κρίμα είναι ότι μέλη νεότερα και παλαιότερα δεν μπορούσαν να παραστούν έγκαιρα για αυτή τη συζήτηση. Καλωσορίζω το έγγραφο αυτό Πιστεύω ότι κάνατε σημαντική πρόοδο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή γι' αυτό. Σίγουρα επιλέξατε αρκετά από τα διαφορετικά θέματα και λεπτομέρειες που είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά. Και καλωσορίζω πραγματικά το γεγονός ότι θα διεξαχθεί ακρόαση. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστια σημασία να εισακούσουμε τους ε, όσους ε, θα εκφέρουν τις απόψεις τους και να διασφαλίσουμε ότι νομοθετώντας θα γνωρίζουμε τις επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας ποιε θα είναι. Και στο μέτρο του εφικτού θα έχουμε προσπαθήσει να ακούσουμε πραγματικά τους εμπλεκόμενους για τις μη στοχευμένες ή τις μη εσκεμμένες επιπτώσεις. Διερωτώ με αν θα υπάρχει ή όχι αν θα ακούσουμε διαφορετικούς από όσους εμπλέκονται στην πραγματική οικονομία, στην ίδια την οικονομία και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να εμβαθύνουμε στα επιχειρήματα για τις επιπτώσεις. Επίσης συνειδητοποιώ τη σημασία της ε, μελέτης επιπτώσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω για το εύρος σχετικά ε, τι πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν όμως και κάποια θέματα που έχω συνειδητοποιήσει που ε, εδώ ουσιαστικά δεν βρίσκονται σε αυτό το έγγραφο επαρκώς. Την τελευταία φορά θα θυμόσαστε ότι μίλησα για τις επιπτώσεις στην ε, υψηλή καινοτομία, καινο, καινοτομία των επιχειρήσεων που με βάση την ατζέντα της Λισαβόνας θα προαγάγουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι η πιο ανταγωνιστική και θα βασίζεται στην τεχνολογία και την καινοτομία. Ε, πήρα χρόνο και αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα ε, σε σχέση με κάποιον που είχε ε, αναμειχθεί με αυτά τα θέματα πριν από κάποια χρόνια. Είναι η δεύτερη ήδη μεγαλύτερη εταιρεία μέσα σε μία δωδεκαετία και έτσι Πρόκειται για τεχνολογία που μέσα σε 12 χρόνια χρησιμοποιούμε σήμερα πια όλοι μας. Ο κύριος αυτός ε, μου επεξήγησε πόσο δύσκολο είναι ήδη σήμερα να έχει κανείς πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου στην Ευρώπη έναντι του τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ για παράδειγμα. Και τα ανέφερε αυτά ως κάποιος που θα ήθελε να προαρθεί η Ευρώπη ως ε, μια οικονομία που θα βασίζεται στις ε, γνώσεις. Όλα αυτά μπορούν να έχουν μη στοχευμένες, μη επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις μας. Σήμερα το πρωί ένα έγγραφο που ακριβώς επεξηγούσε τι γίνεται σε σχέση με τις απαιτήσει για κεφάλαια μέσα σε αυτή την οδηγία και τι αυτά θα μπορούσαν να συνεπάγονται για εκείνους που χρειάζονται τέτοιου είδους κεφάλαια για να ξεκινήσουν τις μικρές επιχειρήσεις τους στην ενακτήρια φάση. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να το θέσω στη διάθεση του εισηγητή. Τα καλωσορίζω τώρα αυτά μέσα σε αυτά τα πλαίσια και μέσα σε αυτόν τον πρόσθετο χρόνο πιστεύω ότι θα έχουμε διασφαλίσει, θα πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή χρονικά όρια ώστε να συζητήσει η βιομηχανία βιομηχανία και να εκφράσει τις απόψεις της με το 1-3 ε, ε, δολαρίων που επενδύονται και που θα μπορούσαν ακριβώς να αναζωογονήσουν τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και έχω περίπου 7 ακόμα αγορητές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Θα σας πω ποιοι είναι. Πρέπει όμως να κλείσει ο κατάλογος ε, των αγορητών. Κλούνκ. Uh, ο Ούντο θέλει να επανέλθει και νομίζω σε σχέση με το σημείο για τη δεύτερη ανάγνωση και εγώ με κάποιες παρατηρήσεις ακόμα μετά το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσουν και θα επανέλθει ο εισηγητής. Αν κάποιος δεν έχει συμπεριληφθεί να μας πει τώρα <clears throat> αν δεν έχει συμπεριληφθεί. Αλλιώς δεν θα προλάβει να παρέμβει μετά. Κλούνκερ τώρα παρακαλώ. Έχω μεγάλα προβλήματα με τα γράμματα εδώ από πλευρά υπαλλήλου γραμματεία. Κλούνκερ, παρακαλώ. Ναι, εντάξει, σα ευχαριστώ λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θερμές ευχαριστίες προς τον εισηγητή για την δουλειά και τον κόπο που έκανε. Σχετικά σύντομος θα είμαι. Θα θε, ήθελα σε μια πτυχή να επικεντρωθώ και να πω ότι αυτό δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα ή δεν αναφέρθηκε κιόλας καθόλου. Είναι απλά οι προβληματικοί ή οι κίνδυνοι που βρίσκονται στο ίδιο το Ταμείο. Είναι δεδηλωμένο στόχο αυτή τη οδηγία οι κίνδυνοι το δυνατόν να αποφεύγονται. Στο μέλλον να αποφεύγονται τέτοιου είδου κίνδυνοι. Όμω έγκυται και βρίσκεται στο ότι και πρέπει αυτό εντονότερα να βρεθεί στο επίκεντρο των προβληματισμών μα στη συλλογή κεφαλαίων αυτών αυτός ο κίνδυνος έγκυται και στο συσσόρευση κεφαλαίου και ο Λόρδος Τέρνερ, ο Άλιστερ Τέρνερ, ο πρόεδρος ε, της ε, ε, Βρετανικής Εποπτικής Αρχής, πρόσφατα μας είπε ότι έχουμε μια διόγκωση αγορών κεφαλαίων και είπε ότι είναι αναγκαίο αυτή η φούσκα να ξεφουσκώσει αυτή η διόγκωση και σε σχέση με το Tobin Stoyer, τον φόρο Tobin ή τον φόρο συναλλαγών που θα, το τέλος συναλλαγών που θα επιβάλλεται, αυτό θα ήταν κάτι ορθό και για την ομάδα τη δική μου της Ενωτικής αριστερά, είναι σημαντικό αυτή η πτυχή να συμπεριληφθεί και να συνεξεταστεί στην έκθεση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι σε αυτή την οδηγία θα δημιουργηθεί μια προϋπόθεση ώστε ένας λογικός τρόπος εφαρμογής αυτού του, στο, του φόρου πανευρωπαϊκά θα έπρεπε να μπορέσει να εισαχθεί. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστούμε. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, Πρόεδρε, τι να σας προσθέσω. Όμως, θα ήθελα απλώς να σας πω ότι εύστοχη νομοθεσία και εύστοχη υποπτία αποτελεί προστιθέμενη αξία όσον αφορά την εναλλακτική μέθοδο επενδυτικών ταμείων στην Ευρώπη, τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Και φυσικά μπορεί να είναι πιο αξιόπιστη η αγορά και επίσης θα μπορέσουμε και αυτόν τον τρόπο να έχουμε καινούργια στάνταρ, να ανέβει ο πύχης γενικά. Να γίνει επομένως μια γενική, σφαιρική ε, εποπτεία και έτσι να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα, τα, τα σωρευτικά αποτελέσματα και από πλευρά λειτουργίες αυτών των οργανισμών θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση των κινδύνων και να προσέξουμε κάτι που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, αυτές τις ε, εξωτερικότητες, τους εξωτερικούς παράγοντες. Γιατί αυτές οι αναλυτικές επενδύσεις δημιουργούν κάποιους κινδύνους ή κάποιες ζημίες που τελικά μετακυλίονται σε όλο τον κόσμο. Άρα, να δούμε τι θα γίνει με την πραγματική οικονομία. Και θα πρέπει ομένω να κάτσει κανείς και να δει τι γίνεται με την αγορά του πετρελαίου, τι γίνεται με την αγορά των ειδών διατροφής. Για να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε των ρυθμίσεων. Επομένω, θα πρέπει κριτήριό μας να είναι η βιωσιμότητα αυτών των οργανισμών και για τα χρέη τους, για τη χρηματοδότηση και να δούμε πώς δεν θα έχουμε στρεβλωτικά αποτελέσματα. Επίσης, όταν μιλάμε για έγκριση λειτουργία, δεν μιλάμε για γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να γίνει πραγματικά διαπίστωση ότι υπάρχει εύρεθμη λειτουργία και ότι υπάρχει εποπτεία και σύνομη λειτουργία. Όποιος επομένως θέλει τέτοιο διαβατήριο ευρωπαϊκό θα πρέπει να υπαχθεί στην ε, ρύθμιση του κοινοτικού δικαίου. Γενικώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντα τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία, τον κύριο εισηγητή Γκοζέ, για την αποσαφήνιση, για την διευκρίνηση που είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή από πλευρά τη εργασία μα όσον αφορά τα διαφορετικά θέματα τα οποία εξετάζουμε. Σε μια χρονική στιγμή όπου η συζήτηση έχει προχωρήσει αρκετά, θα ήθελα απλά και μόνο να κάνω κάποια σχόλια σύντομα Κάποιε παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ισορροπημένο. Η δική μας οδό, η δική μας πορεία πρέπει να στοχεύει σε μια καλύτερη ρύθμιση, βελτίωση των ρυθμίσεων. Δεύτερο, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι αναγκαίο να δούμε τον συντονισμό σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν πολλά θέματα όπου Αζητείτε αυτή η δράση και αυτό είναι μία πτυχή και δεν θα πρέπει να, σε σχέση με τον κίνδυνο να υπάρξει μία ε, πορεία που δεν θα συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα είναι αποτελεσματική. Τρίτον, είναι μία ρύθμιση που πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα. Δηλαδή πρέπει να δει τις επιπτώσεις που τα διαφορετικά ταμεία που εξετάζουμε εδώ, τις επιπτώσεις που έχουν στην ενιαία εσωτερική αγορά. Και κάποια από αυτά τα ταμεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την φερεγγιότητα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης, διεθνού κρίση κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και που δεν ξέρουμε πώ θα τερματιστεί. Τέταρτο, όπως και πριν από λίγο αναφέρθηκε από τον κύριο Γκαρσία Μαργκάλιο, είναι αναγκαίο να δούμε να αντιμετωπίσουμε με ίσο τρόπο, με ίσο τρόπο αλλά και διαφοροποιημένα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα είναι μια πτυχή που αντικειμενικά θα απαιτήσει πολλή δουλειά από πλευρά μα σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει σοβαρά να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία των διαφορετικών ταμείων και να τα εξετάσουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν διαφοροποιημένα και τις διαφορετικές στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν ιδιαίτερα για το θέμα των ίδιων κεφαλαίων την αξιολόγηση των ενεργών κεφαλαίων και την ασφάλεια των μηχανισμών ε, για τις καταθέσεις. Και τέλος επίσης, ε, για να ολοκληρώσω, να πω ότι αυτή είναι μια νομοθετική εργασία που φυσικά πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό που ιστορικά έχουμε στην κοινότητα και να καταλήξουμε σε σχέση με μια ενιαία αντιμετώπιση όσον αφορά τους ε, μηχανισμούς για τις επενδύσεις και για τις αγορές και τα μέσα τα οικονομικά για τις αγορές. Έχουμε πολλά, ε, ε, πολλή δουλειά να κάνουμε για να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον εισηγητή μας που έχει πολύ σημαντικό ρόλο και θέλω να τον ενθαρρύνω στο έργο του. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Λάμπερτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένα σχόλια ε, πρώτον, όσον αφορά το κεφάλαιο κινδύνου, venture capital στην τεχνολογία. Λαμβάνονται υπόψη ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση ε, ως, ε, από venture capital όσον αφορά την τεχνολογία. και βεβαίως οπωσδήποτε σε αυτήν την τεχνολογία και την πράσινη τεχνολογία αυτού του είδους, οπωσδήποτε οι Αμερικανοί μας έχουν ξεπεράσει. Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι ε, διακινδυνεύουν, διακινδυνεύουν, θέτουμε σε κίνδυνο αυτές τις επενδύσεις ε, γιατί, με αυτή την οδηγία, γιατί εδώ έχουμε ένα, μια αγορά η οποία δεν έχει καμία ε, ε, καμία ε, καθοδήγηση κατά κάποιο τρόπο και εγώ λέω ότι ενδεχομένως ακριβώς γιατί έχουμε την δυνατότητα να πάμε σε οποιοδήποτε είδους επένδυση ενδεχομένως τα venture capitals δεν πηγαίνουν στη τεχνολογία αλλά πηγαίνουν σε κεφαλαϊκά προϊόντα ε, δεν θα συμφωνήσετε ενδεχομένως θα πείτε ότι εγώ τώρα το λέω γιατί προέρχομαι αυτή τη βιομηχανία και με ενδιαφέρει. Επίσης κύριε Σμιτ αυτή η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Την ακούω ε, να ε, γίνεται λόγος για αυτήν σε όρους επιτυχημένους. Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε, βεβαίως. Είναι γεγονός ότι εκατομμύρια Βραζιλιάνων, Ινδών, Κινέζων βγήκαν από την ένδια αλλά όμως εάν δούμε την κρίση ε, των τροφίμων, την κρίση ε, του κλίματος, την κρίση των ε, κεφαλαιακών και τραπεζικών προϊόντων, τότε θα καταλάβουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αφρική σαν Ήπειρος, τότε θα καταλάβουμε ότι και αυτό είναι ένας αντίκτυπος ε, του συστήματος. Είναι διαφορετικού είδους αντίκτυπος ε, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Βεβαίως θέλουμε παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά με τις απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα, ε, ε θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν οι τράπεζες βοηθούσαν ε, έτσι ώστε να διευθετείται σωστά το σύστημα, πράγμα που δεν συμβαίνει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υπάρχον σύστημα μπορεί να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, επίσης εγώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμουν στη βιομηχανία και ξέρω ότι το κύριο μέλημα της ε, βιομηχανία είναι, ε, η, ε, είναι η, η μη διακύβευση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μέλων, των stakeholders. δηλαδή αυτό τους απασχολούσε πάντοτε ε, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αρμονία ανάμεσα ε, στα ενδιαφερόμενα μέρη, το κοινωνικό όφελος ε, και τα το, κοινό όφελος. Επομένως, εάν θα πρέπει να, αν θέλετε να συνεχίσουμε έναν διαρκή διάλογο με την βιομηχανία, βεβαίως συμφωνώ μαζί σας. Εάν λέτε ότι πρέπει να σταματήσει ο διάλογος με το κοινό, ο διάλογος με τους εκλογείς μας, ε, τότε ε, εντάξει δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ε, γιατί μπορεί να λέτε εσείς ότι οι εκλογές τελείωσαν αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τους ακούσουμε τουλάχιστον όσο θα ακούσουμε και τη βιομηχανία. Thank Ο κύριος Κάρας παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισηγητά, για αυτό το θέμα θέλω να πω ότι χαιρόμαστε για το ότι είναι ο εισηγητής ο Γκοζέσε Είναι μεγάλη ελπίδα, αλλά χωρίς εμάς δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα. Γι' αυτό θα έπρεπε το κλίμα αυτής της συνεργασίας, η ατμόσφαιρα αυτή να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια του έτους και της εργασίας συνολικά. Κάποια πράγματα είναι σημαντικά εδώ. Το πρώτο είναι την οδηγία αυτή θα την χρειαζόμαστε ακόμα και χωρίς την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Θα την χρειαζόμαστε δηλαδή ούτως ή άλλως, ακόμα και χωρίς κρίση. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται μόνο ως επίπτωση της χρηματοοικονομικής ε, κρίσης να συζητηθεί και να αξιολογηθεί. Εντάξει, διότι κατά τα άλλα θα καταλήγαμε σε εσφαλμένα, σε λανθασμένα συμπεράσματα για την πραγματιστική προσέγγιση του τι θα πρέπει να ρυθμιστεί. Υπάρχει κοινό, ε, κενό ρύθμισης εδώ που πρέπει να καλυφθεί και χωρίς την κρίση θα έπρεπε να ρυθμιστεί λοιπόν. Δεύτερο στοιχείο. Και εδώ πάλι και στην Επιτροπή μας. Πολλοί στη συζήτηση με τους Αμερικανούς θεώρησαν ότι τα επενδυτικά κεφάλαια investment funds δεν είναι το αίτιο της κρίσης. Αν δεν είναι λοιπόν το αίτιο της κρίσης, ε, τότε αυτή την οδηγία θα έπρεπε πολύ πιο νυφάλια και πολύ ευρύτερα, με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής να την ε, εξετάσουμε. Μετά το όνομα, τίτλος. Έχουμε κεφάλαια που λένε ότι δεν θεωρούμε ότι είμαστε εναλλακτική λύση στα επενδυτικά κεφάλαια, αλλά εντασσόμαστε σε αυτή την οδηγία αν παραμείνει ο τίτλος ως έχει αναλύωτος. Πιστεύετε ότι εδώ κάποιο μειονέκτημα μπορεί να ε, υπάρξει ως επίπτωση για κάποιους που εμπλέκονται. Και τώρα πρέπει νομίζω τον τίτλο, το όνομα να το συζητήσουμε. Προσωρινά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν αφορούν όλα τα funds, ε, τα κεφάλαια αυτά. Δεν είναι ο κάθε ένας, το κάθε ταμείο από αυτή τη δραστηριότητα μια εναλλακτική ε, ε, επενδυτική δραστηριότητα. Έχουμε κεφάλαια που αποκλειστικά δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και όχι διασυνοριακά. Και εδώ πάλι τίθεται το ερώτημα. Θα διαφοροποιήσουμε στη ρύθμιση ναι ή όχι τη σχετική αυτή δραστηριότητα. Το τέταρτο σημείο παρατήρηση Μέχρι τώρα μόνο οι διοικητικέ αρχές ε, ε, καλύπτονται. Θα έπρεπε και τα ίδια τα ταμεία, τα ίδια τα κεφάλαια να καλύπτονται, όχι μόνο η διαχείριση, η διοίκησή τους. Έχουμε διαφορετικά κεφάλαια που εντάσσονται όλα σε αυτή την οδηγία. Θέλουμε όμως όλα αυτά τα κεφάλαια, όλα αυτά τα ταμεία σε αυτή την ε, οδηγία, παρότι έχουν διαφορές στη δραστηριότητά τους ενιαία να τα αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται εδώ συστημική προσέγγιση. Χρειάζονται αρχέ για τα κεφάλαια και τους ε, διαχειριστές, τους διοικητές που θα ισχύουν για όλους βέβαια αλλά χρειαζόμαστε εξειδικευμένες, εξειδικευμένες ρυθμίσεις που θα αφορούν τις ιδιομορφίες ε, των κεφαλαίων αυτών εκάστοτε και να δούμε αν θα τα ρυθμίσουμε εδώ πανευρωπαϊκά ή αν οι, αυτο, ε, οι μηχανισμοί αυτορύθμισης από πλευράς των κεφαλαίων των ταμείων αυτών επαρκούν για παράδειγμα σε περιπτώσεις που μόνο σε ένα κράτος δραστηριοποιούνται και όχι διασυνοριακά η αρχή ένας, μία ρύθμιση για όλους, για τα ταμεία, θα πρέπει να καλύπτει τα κοινά του στοιχεία και μετά με διαφορετικό τρόπο να προβούμε στη ρύθμιση των εξειδικευμένων θεμάτων που δεν επιτρέπεται ισοπεδωτικά να αντιμετωπίζονται. Τελευταία μου παρατήρηση αφορά το χρονοδιάγραμμα. Όλε Σμιτ, Νομίζω γι' αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια αντιπαράθεση. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να το πω έτσι, αν δεν είναι ε, δυνατόν να ολοκληρωθούν όλα αυτά, ε, αν αυτά ολοκληρωθούν έγκαιρα δεν θα καταλήξουμε σε τριμερείς διαλόγους. Και για τη ρύθμιση αυτή de facto να δούμε ότι σε σχέση με, την, το Συμβούλιο και την ε, κοινή θέση θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Εδώ οι δυσκολίες στο Συμβούλιο είναι πολύ μεγαλύτερες, διότι και η προσέγγιση από πλευρά τους είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με εμά με την Ευρωβουλή αν αυτή την φάση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μπορούμε να, τις, ε, να την ε, απαλείψουμε, αν ε, ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Αν δεν φτάσουν σε αυτό το σημείο δεν θα καταλήξουμε σε τριμερείς διαλόγους αλλά αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν θα κάνουμε την πρώτη ανάγνωση εμείς και δεν θα περιμένουμε τριμερείς διαλόγους. Ευχαριστώ. Right, Ο κύριος ε, Τρεμός έχει ζητήσει το λόγο. Μόνο ένα λεφτάκι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω αυτό το λεπτάκι για να σας πω κάτι. Ε, άκουσα σήμερα το πρωί πολλούς ανθρώπους να ζητούν περισσότερο έλεγχο, περισσότερη υποπτία, περισσότερη νομοθεσία. Και εγώ τώρα επιφυλάσσομαι σε σχέση με τις αιτίες της κρίσης έχετε μήπως κατά νου της, την τραπεζική κρίση του, του, του, του, τέλους του 19ου αιώνα. Μα τότε δεν είχαμε κάποια κεντρική τράπεζα, κρατική, με μονοπόλιο, κοπής νομίσματος. Σήμερα έχουμε τις κεντρικές τράπεζες. Οπότε και γι' αυτό τότε, ας πούμε στη είπα, είχαμε πολύ περισσότερες τραπεζικές κρίσεις από ό,τι σήμερα γι' αυτό το λόγο. Οπότε, και η κρατική παρέμβαση και οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη αποτελούν τμήμα των αιτιών της κρίσης. Ας πούμε, την, ε, την, την τεχνητή διαμόρφωση από τις δημόσιες τράπεζες των επιτοκίων. Επί πολλά χρόνια τεχνητά καθοριζόντουσαν χαμηλά επιτόκια και έτσι επομένως είχαμε κάποιο είδους ε, άνθηση της αγοράς των πιστώσεων που ήταν τεχνητή, οπότε και οδηγηθήκαμε σε, σε, σε υπερχρέωση και σε στροφλωτικά φαινόμενα. Οπότε, σας παραμένω σε αυτό που είπε ο Όλε Σμιτ. Οπότε, να κάτσουμε να ξανασκεφτούμε τα όσα μα είπαν όσοι θέλουν περισσότερη παρέμβαση. για πετε μου, του φύλακε ποιο του θα του φυλάει. Θα του δώσουν περισσότερες εξουσίε τώρα. Μπούλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον συνάδελφο Όλε Σμιτ. Ο συνάδελφος Όλε Σμιτ κατά την τελευταία συνεδρίαση και άδικα όπως βλέπω, ήταν άδικος μαζί μου όταν είχαμε τα θέματα της ε, ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν έγινε κατανόηση από, δεν έγινε κατανοητή η δική μου προσέγγιση από πλευρά του αλλά δεν μνησεί κακό και έχει, δίνω δίκιο όσον αφορά την προσέγγιση ως ιδέα πρέπει πρόεδρε κανονικά από διαδικασία συναπόφασης με δύο γύρους να ξεκινήσουμε έχει δίκιο όταν λέει ότι εμείς ως νομοθέτης, ως νομοθέτης πρέπει να κάνουμε σωστά το έργο μας. Και εμείς το βλέπουμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και αν ο Ότμαρ Καράς έχει εδώ μια παρατήρηση που και έχει δίκιο και πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε το Συμβούλιο τότε αυτή η κατάσταση δημιουργείται ακριβώς επειδή με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση συνειδητά καταλήγουμε σε μια διαδικασία δύο γύρων όταν την προσεγγίζουμε έτσι. Αλλά μην δώσουμε λάθος μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι ευθύ εξ αρχή εκινούμε από μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να βοηθήσει. Δεν βοηθά και τον εισηγητή στην πολύ δύσκολη δουλειά του. Και συμφωνώ λοιπόν με αυτή την παρατήρηση που ε, εξέφρασε ο Σμιτ. Σας ευχαριστώ. Λέγει πρόεδρος. Έχω αρκε... Υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις, ε, ε, διευκρινιστικές περισσότερο που θα έπρεπε να κάνω και όχι τόσο επί της ε, ουσίας ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω φυσικά ότι ξεκινήσαμε νωρίς επειδή διακόπτη πρόεδρος. Όταν τελειώσει ο Ρόμπερτ θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη συζήτηση νωρίς, πρώιμα. Κάποια μέλη αυτό το, τα εξέπληξε, διότι ήταν συντομότερα τα προηγούμενα σημεία από ό,τι αναμενόταν. Αν κάποιοι έχασαν λοιπόν τις πρώτες παρεμβάσεις που ήταν ουσιαστικές, ιδιαίτερα των σχεδόν εισηγητών και του κυρίου Μπούλμαν τις παρατηρήσεις, και από πλευράς του κυρίου Καμάλ και άλλων συναδέφων για παράδειγμα θα σας στείλουμε την, ε, την συνεκτική αυτή αναφορά όσον αφορά το αρχείο μας ε, από το διαδίκτυο ε, όπου διαχαιόταν αυτή η συζήτηση και μπορεί να επιλέξετε λοιπόν τις παρατηρήσεις που σας ενδιαφέρουν και σε σχέση και με τις ε, παρεμβάσεις από πλευράς ε, ε, των συναδέφων όσον αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επίσης, όσον αφορά τώρα το χρονικό, την χρονική συγκυρία, είναι σημαντικό τα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα ανοιχτό πλαίσιο και αποτελεσματικά. Είχα αναφέρει στις 2 Σεπτεμβρίου αν θέλαμε να, πάμε, να ακολουθήσουμε την προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης και υπήρξαν κάποιες ανησυχίες και υπήρξε υποστήριξη για μια συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Είναι δουλειά της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να λάβει μια τέτοια απόφαση. Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι εύκολο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση χωρίς ε, πρώτα να έχουμε προχωρήσει κάπως. Πρέπει να παραμείνουμε σε ένα ανοιχτό πλαίσιο θα έλεγα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υπενθυμίσω στον εισηγητή ότι εμείς είχαμε μια εμπειρία με την οδηγία περιπληρωμών όπου έπρεπε πολλές τροπολογίες και αναδιατυπώσεις, αναδιατυπωτικό έργο να γίνει. Και αυτό σε σχέση με ένα έγγραφο τριών στυλών δημιούργησε προβλήματα. Εσείς σας το εισηγητής και ήταν δυσχερές αυτό το εγχείρημα σίγουρα. Έχουμε λοιπόν κάποιο βίωμα σχετικά, κάποια πείρα, γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε εξοικειωθεί με αυτά. Θα ήθελα να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παράσει ένα πίνακα για τις, ε, δια, την διασύνδεση αυτού του θέματος με άλλες διαφορετικές οδηγίες και με την, ε, τις επικαλύψεις όσον αφορά την οδηγία για τις ε, χρηματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όσον αφορά και την αποφυγή της, του δεσπόζοντος ρόλου και της, του καταχρηστικού ρόλου και την οδηγία για ρευστότητα 2 και σίγουρα όλα αυτά και με ένα link με τις διάφορες οδηγίες όσον αφορά λογιστικά θέματα και απαιτήσει και την τρέχουσα ε, ρύθμιση όσον αφορά τις εποπτικές αρχές, τη δομή τους, τη διάρθρωσή τους για την επιτήρηση. Έτσι λοιπόν μια σαφής ε, ε, επεξήγηση για τις αμοιβέ επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν. Τώρα, για, τις, για την αξιολόγηση επιπτώσεων, δύο θα έχουμε. Μία που θα είναι έτοιμη κατά τα τέλη Οκτωβρίου και μία δεύτερη που θα είναι έτοιμη κατά τα τέλη Νοεμβρίου και ε, θα δούμε περαιτέρω το θέμα αυτό για το εύρος και μέσα ε, στο πλαίσιο ε, στο οποίο πρέπει να τηρηθούμε να δούμε κατά πόσον μπορεί αυτό να τηρηθεί και να καλύψουμε τα κενά τα οποία θα υπολείπουν μετά στη συνέχεια. Αυτό είναι το, η κυριότερη προσέγγιση μας. Για το web streaming το είπα ήδη πιο πριν και φυσικά επανερχόμαστε κάποιοι από εμάς όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα τεκτενόμενα και τον, την ανάγκη διεθνώς να υπάρξει ένας συντονισμός και αυτό έχει ήδη αναφερθεί σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ η ίδια για την ιδέα αυτή που εισήχθη από πλευράς Κλίντ ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό ποιοτικά, με αναβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά τις προδιαγραφές. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Και εν τέλει, σε σχέση με τις νομικές υπηρεσίες ε, της, ε, του Ευρωκοινοβουλίου και της ε, κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής, θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει σε ένα θέμα του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και για τις, τους όρους και προϋποθέσεις αμοιβαιότητας. Διότι έχοντας δει αυτό σε σχέση με άλλες οδηγίες και σε σχέση με το solvency του την οδηγία για τη, τη ρευστότητα 2 οι ε, νομομαθείς μας είπαν ότι θα έπρεπε να ε, δούμε το θέμα της ε, αμοιβαιότητας και των ε, διατάξεων για τις, ε, την, αμοι, την αμοιβαιότητα ε, θα ήθελε η Επιτροπή να απαντήσει επ' αυτού. Πρώτα θα λάβει τον λόγο η Προεδρία, μετά θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά ο εισηγητής. Έχουμε περίπου ένα τετατάκι 20 λεπτά συνολικά για να τα καταφέρουμε. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ήταν όλα τα όσα άκουσα στην συζήτηση σήμερα. Συγγνώμη, γιατί και εγώ έχασα την αρχή της συζήτησης. Πάντως, σε αυτή τη φάση, το μόνο που πρέπει να σας πω είναι για το οποίο ελέγχθη από κάποιο βουλευτή, όσον αφορά την διαφάνεια μεταξύ ημών και ημών ότι σκοπεύουμε να αποκτήσουμε τέτοια διαφάνεια. Ακόμα και αν δεν θα έχουμε την Προεδρία όταν ολοκληρωθεί ε, αυτό το θέμα. Οπότε, θα σας πω πως ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα εδώ μας εξήγησε ο εισηγητής, πάρα πολλά από όσα είπε ε, ισχύουν Ελπίζω επομένω να τα πάμε πάρα πολύ καλά και να επιτυχημένη συνεργασία μα. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έγγραφό σα μπορούμε να το διανύμουμε. Έχουμε όλα τα επιμέρου θέματα σε κάποιο έγγραφο, το οποίο όντω δεν είναι βεβαιωμένο και προ για δημόσια χρήση. Μα μπορείτε να το βρείτε στο website. Αυτό υπάρχει μόνο στο website. Αυτό. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει λόγο. ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να αρχίσω κάτι θετικό, ότι δηλαδή τελικά, να, που βρέθηκε κάτι που είναι κοινό προνομαστής. Όλοι χάσαμε την αρχή των ε, των Και αυτό είναι υπομένως ένα κοινό σημείο. Να, κάτι λοιπόν, πάρα πολύ Και άρα, ας κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε στο web stream ε, τις αρχικές εισηγήσεις. Τώρα, για να δούμε τώρα κάποια άλλα πιο ελαφρά θέματα. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή την οποία συνέταξε ο κύριος Γκοζές οπωσδήποτε αναδεικνύει τα πιο βασικά θέματα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Μα δείχνει την κατεύθυνση που θα πει, πρέπει να βαδίσουμε για να διεκπαιρεώσουμε το θέμα και θα σας σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Και έτσι νομίζω ότι θα απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί και μεταξύ των άλλων και εσείς Πρόεδρε θέλετε να σας τα εξηγήσουμε. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, όσον αφορά την εμβέλειά της, θεωρούμε ότι αυτή η προτινόμενη από εμάς είναι η πιο σωστή προσέγγιση. Για λόγους πρακτικούς ή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο να κάτσουμε να καλύψουμε νομικά όλα τα διαφορετικά μοντέλα των σχετικών επιχειρήσεων. Να κάτσουμε, δηλαδή, ή να κάτσουμε να εξαιρέσουμε τη ρύθμιση κάποιου τύπου ε, τέτοιων ε, επιχειρήσεων. Όμω, αλλά και από πλευρά πολιτική, αυτό είναι ο πιο σωστό τρόπο να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα όσα ε, αποφασίστηκαν από το G20 όπως είπε κάποιος βουλευτής. Άρα, θέλουμε να είναι μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια του νομοθετήματος για να καλύψει όσο γίνεται περισσότερους τύπους επιχειρήσεων. Βεβαίως, έχουμε πιστεί ότι στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες για να προσαρμοστούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες κάποιων συγκεκριμένων μορφών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να πέσουμε στην παγίδα του να κάτσουμε και να δώσουμε κάποιους ορισμούς, γιατί τότε θα ξαναέχουμε το γνωστό πρόβλημα. Να δούμε ομένως τι δραστηριότητα να πτήσει το κάθε μοντέλο, τι χαρακτηριστικά έχει και Όπω περιέφερε να κάνουμε περισσότερο. να κάτσουμε μέρο να, να, να, να δούμε σε τι βαθμό θα πρέπει να γίνει κάποια διαφοροποίηση, οπότε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό σκοπό, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε κάποια λογική, αναλογική, δόκιμη νομοθεσία. Το αυτό το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή τη σχέση αυτού του νομοθετήματος με τα υπόλοιπα που ήδη ισχύουν για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ξέρουμε ότι εκ πρώτης όψεως ίσως υπάρχει κάποιος κίνδυνος επικάλυψης. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την επικάλυψη όσο γίνεται περισσότερο. Θα προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την υπάρχουσα ε, νομοθεσία με αυτήν την πρόταση. Να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδου ε, συνέργεια και όχι επικάλυψη. Με βάση αυτού του εγγράφου που υποβιβλήθηκε στο Συμβούλιο. Και έτσι να μπορέσουν σαν το Συμβουλίου να έχουν κάποια εγγραφή εργασία και να συνεργαστούμε. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που ανακύπτουν σωστά όσον αφορά αυτή την αναγκηρύθμιση. Να μην έχουμε κενά παραθυράκια δηλαδή, στην ρύθμιση. Ρίξτε μια ματιά και πέστε μα, νομίζουμε ότι το εγγραφό μα πάντω σα δίνει κάποιε απαντήσει Τώρα, η σχέση, η σχέση με την αρχιτεκτονική των υποπτικών αρχών. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση μάλλον είναι πρόημο να κάτσουμε και να απασχοληθούμε με αυτό. Βεβαίω και θα πρέπει να μα προβληματίσει, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπω ε, πρόημα σε σχέση με την πρόταση της ε, Κομισιόν που ήδη έχει πρώτα υποβληθεί. Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Δύσκολο όμως να κάτσουμε να λάβουμε υπόψη όλους του παράγοντες σε αυτή τη φάση. Κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ένας νέος οργανισμός μπορεί να επιλύσει κάποια αυτά τα προβλήματα που ετέθησαν. Για τρίτος χώρας κάτι τελευταίο. Είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα αυτό, βέβαια δεν μπορεί να λυθεί σήμερα. Όμω με την ευκαιρία, σε δύο λεπτά για να σα ε, πω ποιε είναι οι προθέσει μα. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά τουλάχιστον σε εξηγήσω γιατί θεωρούμε ότι οι προθέσει μα δεν είναι καθόλου το να καταλήξουμε σε μέτρα προστατευτικά. είχαμε ως πρότυπο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κάτι το οποίο σε αυτό το τομέα δεν είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά για άλλου είδους ε, νομοθεσίες συνηθίζεται πάρα πολύ. Έχουμε μόνο κάποιους κανόνες για τους διαχειριστές που δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που φυσικά η δράση τους έχει επιπτώσει στα ταμεία. Αυτός είναι πάνω στο στόχο της ρύθμισης. Θέλουμε επομένως για αυτούς τους διαχειριστές να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την προσβασιμότητα και στους διαχειριστές τρίτων χωρών. Όμως, υπό τον όρο της ισοδυναμίας ή αμοιβαιότητας. Υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει του διαχειριστέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και για αυτού που προέρχονται από τρίτες χώρε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα με την οδηγία, αλλά μπορεί να γίνει με τον έλεγχο αμοιβαιότητα οτιμίας, ισοδυναμία. Αυτή είναι η πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει όμω και οι δικοί μα και οι ξένοι να μπορούν επί τη βάση της ισοτιμίας να ενεργούν. και με αυτό το πανευρωπαϊκό διαβατήριο να μπορούν να ωφεληθούν και οι παράγοντες των χωρών και οι κοινοτικοί. Κατηγορηθήκαμε επομένω ότι πρόθουμε προστατευτισμό. Αλλά ε, μας παρέχει ανακούφιση το ότι από άλλους θεωρήθηκε προβολικά φιλελεύθερη, ένας δούριος ύπος. Επομένως αυτό το πνεύμα μας διαπνέει και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τελικά μάλλον ισορροπημένα τα βλέπουμε. Ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας και όπως συνεχθήκαμε μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε σε συνεργασία και με εσάς αλλά και με το Συμβούλιο. Μπορείτε να μας υπολογίζετε. Και έτσι να πετύχουμε τον κοινό στόχο. Πρόεδρος. Ενδεχομένως ε, θα σας στείλουμε τα σχόλια της ε, νομικής ε, υπηρεσίας. Θα σας το στείλουμε για να το σχολιάσετε και να μας στείλετε ξανά την απάντησή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καμιά φορά στο Κοινοβούλιο ε, συζητούμε, χρησιμοποιούμε εμφατικές λέξεις, πομπόδεις λέξεις. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ήταν πραγματικά πλούσια αυτή η συζήτηση και ότι όλοι κατάφεραν να ε, πάρουν το λόγο και αυτό είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό. Τώρα, θα ήθελα να σας πω σε όλους όσους ανησύχησαν που έχασαν την αρχική μου παρέμβαση ότι είπα ελάχιστα πράγματα, δεν θα περάσετε πολλή ώρα για να το δείτε ηλεκτρονικά. Ε, είπα ότι από τη στιγμή που υπήρχε το γραπτό κείμενο ε, δεν υπήρχε λόγος να ξαναπώ αυτά που είχαν ήδη διαβάσει και του περίμενα τα δικά του σχόλια. Λαμβάνω υπόψη μόνο τα σχόλια που άκουσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερω τους σκιώδει συγητές για την εργασία τους, για την προσπάθειά τους. βεβαίω έχω έρθει ήδη σε επαφή μαζί τους και είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε όμου να βρούμε απαντήσεις στις ε, πολυπληθείς ερωτήσεις και ε, θα ήθελα να πω στον κύριο Σμιτ ότι ακούω όλους όσους έρχονται να μου μιλήσουν ε, και πραγματικά τούτο το διάστημα, τούτη την περίοδο ε, δέχομαι πάρα πολλούς επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ακρόαση που προετοιμάζεται κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν ε, οι μελέτες ε, επιπτώσεων, ένα σύνολο πραγμάτων. Γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Πολύ σύντομα να εξάγω κάποια συμπεράσματα, και κάποιες κεντρικέ ιδέες. Πρώτον, μεγάλη πλειοψηφία επί της ιδέας ότι χρειάζεται διακανονισμός. Ε, και νομίζω ότι όλοι πολύ σοβαρά λένε ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε αυτό το έγγραφο, να το στείλουμε στον κάθε των αχρήστων. Επίσης, ε, ε, ορθολογικός διακανονισμός, ορθολογική ρύθμιση που θα είναι και αποτελεσματική ρύθμιση. Και η πρόταση που μας υποβάλλεται ε, χρειάζεται αποσαφήνιση και ορισμών και κανόνων και διαφοροποίηση των κανόνων έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση και η πληθώρα των εργαλείων που καλύπτονται από το ευρύ φάσμα εφαρμογή τη οδηγία. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά πράγματα τα οποία εξάγω ω συμπεράσματα από τι ε, πολύ ορθέ τοποθετήσει ε, των συναδέλφων. Ε, και επ' αυτών των στοιχείων θα προσπαθήσουμε να ξαναδούμε το κείμενο. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, έχουμε μεγάλη εμπειρία κειμένων που χρειάζονται χτένισμα και βεβαίω δεν ήταν πολύ λυπηρή η θέση του Κοινοβουλίου αν η Κομισιόν μα έδινε εξαιρετικά κείμενα που δεν θα χρειάζονται καμία διόρθωση. Νομίζω ότι και οι συγητέ και οι σκιώδει συγητέ και όλοι οι υπόλοιποι και οι Κομισιόν ε, βάζουν ε, το λιθαράκι του στο οικοδόμημα. Ε, και όπω είπε και ο φίλο μου ο Ρομπέρ, η Επιτροπή προτείνει και το Κοινοβούλιο αποφασίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει